Καλημέρα σε όλους σας. Ε, θα κηρύξω την έναξη συνεδρίασης γιατί έχω μερικές ανακοινώσεις. Πρώτον, έγκριση της μερίσιας διάταξης. Δεν διαφωνεί κανείς. Συνεχίσω. Ανακοινώσεις δεν θα τις ακούσει κανείς γιατί δεν είναι εδώ, αλλά θα τις κάνω. Η Επιτροπή μας ψήφισε σε 7 Μαρτίου 2011 την έκθεση για τις χρηματαγορές και το short selling, τις ακάλυπτες ε, πωλήσει και στη συνέχεια ο εισηγητής δήλωσε την πρόθεσή του να αρχίσει διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για το θέμα αυτό που είναι και προτεραιότητα της Επιτροπές μας. Ε, σύμφωνα με τις στάνταρ διαδικασίες η εντολή διαπραγμάτευσης θα ψηφιστεί και θα συμμετέχουν στη διαλλαγή η Πρόεδρος, ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές. Ξέρω ότι δεν έχει διαφωνήσει κανείς, δεν υπάρχει αντίρρηση και θα συνεχίσουμε έτσι. Επίσης, στις 16 Μαρτίου ψηφίσαμε την έκθεση για τη διασυνοριακή εφαρμογή του Eurocast by Road. Η συγκήτρια επίση θέλει να ε, το ε, συμφωνήσει σε πρώτη ανάγνωση και σύμφωνα με τις τρέχουσε διαδικασίες η διαπραγματευτική εντολή θα είναι η έκθεση όπως ψηφίστηκε και θα συμμετέχουν στη συνδιαλλαγή πρόεδρος, εισηγήτρια και σκιώδης εισηγητές. Ξέρω επίσης ότι δεν έχει ε, αντίρρηση κανένας και σε αυτό το θέμα και θα ακολουθήσουμε την διαδικασία. Και τέλος, η Επιτροπή μας στις 22 Μαρτίου θα ψηφίσει, αύριο δηλαδή, την έκθεση για την ε, επιπλέον ε, εποπτεία των χρηματοοικονομικών ομίλων κτλ. Για την εκτελεστική οδηγία θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της αυριανής απογευματινής ψηφοφορίας θα ψηφίσουμε και για το διορισμό των ε, υποψηφίων που έχουν επιλεγεί για την ε, αρχή εποπτείας των χρωματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό είναι λοιπόν και το δύο τέλος των ανακοινώσεων, το τρία αναβλήθηκε και μπορούμε να περάσουμε στο χρονοδιάγραμμά μας το ενδεικτικό νομισματικός διάλογος με τον κύριο Τρισέ. Θα βγω έξω να δω τους συναδέλφους που περιμένουν τον κύριο Τρισέ και απέφυγαν να ακούσουν τις ανακοινώσεις. Okay, um, Σας ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον Jean-Claude Trichet, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τον νομισματικό διάλογο. Όπως θα γνωρίζετε πολλοί από εσά, επί μία ώρα συζητάει μαζί μας ε, λεπτομερώς ε, διάφορα ζητήματα της δέσμης ε, μέτρου για την οικονομική διακυβέρνηση και με πολύ μεγάλο θάρρος έρχεται αμέσως χωρίς διάλειμμα να συνεχίσει τις συζητήσεις στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τρισέ. Θα ακούσουμε πρώτα τον Ζαν Κλοντ και στη συνέχεια ε, τη συνήθη συζήτηση θα έχουμε. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very, very much indeed, Madam Chair. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτές. Όπως κατ' επανάληψη στο παρελθόν, η πάγια συνάντησή μας γίνεται σε έκτακτους καιρούς με τραγικές εξελίξεις στην ε, η Ιαπωνία με το θλιβερό γεγονός ε, απώλειας ανθρώπινων ζώων. Εδώ στην Ευρώπη σίγουρα η ακρόση πέφτει ε, σε μια χρονική στιγμή ανάμεσα σε δύο συναντήσει των Πρωθυπουργών Κρατών και επικεφαλή κυβερνήσεων και το ΕΚΟΦΗΝ και με σημαντικέ αποφάσει για την οικονομική διακυβέρνηση και πριν έρθω στι οικονομικέ προοπτικέ και τα θέματα για σήμερα, θα ήθελα να σα πω δύο λόγια για την μεταρρύθμιση όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Όπω ξέρετε, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε μια γενική μέθοδο προσέγγιση στο θέμα αυτό αυτή η μέθοδος αφορά διάφορες βελτιώσεις. Ωστόσο, πολλές από τις σημαντικές προτάσεις για να ενισχυθεί αρκετά το πλαίσιο διακυβέρνησης ακόμα δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αυτό απαιτείται για να διδαχθούμε πλήρως από την κρίση, γιατί οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μας που ενδιαφέρει το, το μέλλον μακροπρόθεσμα ζητούν από τις αρχές να κάνουν ό,τι απαιτείται έτσι ώστε να αποφευθεί η επανάληψη των εξελίξεων που ζήσαμε τα τελευταία 7 χρόνια. Έτσι, με βάση ε, μια πρόσφατη σφημομέτρηση του Ευρωβαρόμετρου, περίπου το 80% των πολιτών στις χώρες της Ευρωζώνης θεωρούν ότι ένας πιο μεγάλος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή μια αποτελεσματική και αποδοτική διακυβέρνηση, απαιτείται για να καταπολεμηθεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Πριν από 10 μέρες, τα κράτη-μέλη έκαναν μια ε, δήλωση σχετικά με την ε, ενδυναμωμένη συνεργασία των οικονομικών πολιτικών στον Ευρωχώρο. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε πολλά σημεία στο περιεχόμενό της των έξι νομοσχεδίων που έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή. Και αντί να αφήσουμε αυτή τη ε, δήλωση εκ να υπάρχει, θα ήταν πολύ καλύτερα να εξετάσουμε τα κεντρικά τη και να τα εντάξουμε στην σημερινή νομοθετική διαδικασία. Αυτό θα βοηθούσε να αποκτήσει καλύτερη αξιοπιστία αυτή η δήλωση προθέσεων. Let me turn to... Και τώρα συνεχίζω στα αγγλικά. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στι οικονομικέ και νομισματικέ εξελίξει από την τελευταία μα συνάντηση τον περασμένο Νοέμβριο. Θα ασχοληθώ κυρίω με την ανάλυση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ε, συνεδρίασή του της 3ης Μαρτίου. Ε, νέες πληροφορίες επιβεβαίωσαν την άποψή μας ότι η κίνηση προς οικονομική δραστηριότητα παραμένει θετική και προσδοκούμε η οικονομία να ωφεληθεί περαιτέρω από την συνεχιζόμενη ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία. Και η νομισματική μας πολιτική, όπως και τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν για την λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όσον αφορά τι εξελίξει στι τιμέ, ο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη αυξάνεται. Το Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,4%, τον Ιανουάριο ήταν 2,3%. Αυτή η αύξηση σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών. Ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις σε τιμές της ενέργειας που οδήγησαν σε ανωδική πίεση τις τιμές στις πρώτες φάσεις της διαδικασίας παραγωγής. Είναι ιδιαίτερα σημασία σε αυτή τη στιγμή να αποφύγουμε η πρόσφατη αύξηση στον πληθωρισμό να μετατραπεί σε δευτερεύοντα αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη μέσω της, ε, του καθορισμού τιμών ή ψηλότερου μισθούς, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα. Κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης ε, Μαρτίου, η κίνδυνοι για την προοπτική όσον αφορά τις τιμές ε, κινούνται ανωδικά, οι τιμέ των πρώτων υλών μπορεί να αυξηθούν περισσότερο από ό,τι περιμένουμε. Επίση, οι έμεση φόροι, οι διοικητικέ τιμέ επίση μπορεί να αποδειχθούν ψηλότερε, επειδή υπάρχει ανάγκη για οικονομική εξυγίανση για τα επόμενα χρόνια. Τέλο, η ανάκαμψη στη δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ε, οδηγήσει σε πιο μεγάλε εσωτερικέ πιέσει των τιμών. Όσον αφορά την μελλοντική νομισματική μα πολιτική, δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που είπα εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου επί τη ευκαιρία της τελευταίας ε, συνάντησής μας στις αρχές Μαρτίου. Όσον αφορά τις ε, πράξεις για τη ρευσότητα, το Διοικητικό Συμβουλίο αποφάσισε ε, να το κάνει στο δεύτερο τρίμηνο του 2011 με τις ίδιες συνθήκες και όρους όπως και το πρώτο τρίμηνο του 2011. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε τις ίδιες διαδικασίες με σταθερό συντελεστή για προσφορές με πλήρη παραχώρηση σε όλες τις πράξεις επαναχρηματοδότησης τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, θα έρθω σε κάτι που μου ζητήσετε ειδικά να συζητήσω και θα αρχίσω με το εθνικό χρέος. Τονίζω για μια φορά και ακόμα ότι ο σωστός τρόπος να αποφύγουμε τον κίνδυνο κρίσεων εθνικού χρέους στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι με υγιή, εθνικές, υγιείς εθνικές μακροοικονομικές πολιτικές και ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι ένας μηχανισμός διαχείρισης της κρίσης μόνιμος θα ήταν χρήσιμος. Από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθορισμός ενός τέτοιου μηχανισμού είναι ουσιώδης προκειμένου να συμβάλλει θετικά στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα να τονίσω τα εξή δύο τινά. Πρώτον, ο μηχανισμός σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποδυναμώσει τα κίνητρα για υγιή, φορολογική και μακροοικονομική πολιτική που ακολουθούν όλα τα κράτη-μέλη. Ειδικά δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τα κίνητρα για ε, ε φορολογική και μακροοικονομική προσαρμογή από τις ενδια... συγκεκριμένες ενδιαφερόμενες χώρες, αποφεύγοντας τον λεγόμενο ηθικό κίνδυνο. Δεύτερον, επειδή η Ευρωζώνη χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό οικονομική και χρηματοπιστωτική ενοποίηση μεταξύ των κρατών, ο μηχανισμό θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει ε, πολλά εργαλεία που θα είναι αποτελεσματικά ώστε να εμποδιστεί η, ε, κατά κάποιο τρόπο η μόλυνση που μπορεί να περάσει ε, όσον αφορά την ε, αστάθεια της αγοράς από χώρα σε χώρα. Επίσης θα πρέπει τα διάφορα κονδύλια και ταμεία να χρησιμοποιούνται με σόφρονο τρόπο. Η παρεμβάση στη δευτερογενή αγορά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά τη θεσμική μέθοδο, προκειμένου να συσταθεί αυτός ο μηχανισμός ESM, η Κεντρική Τράπεζα όπως και το Ευρωκοινοβούλιο, είναι υπέρ της πιο μεγάλης δυνατής πρόσβασης χρήσης της κοινοτικής μεθόδου. Έχουμε την εμπειρία και μπορεί ο μηχανισμός αυτός να γίνει ένας μηχανισμός της Ένωσης την κατάλληλη χρονική στιγμή. Στο μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα ενθαρρύνει την αξιολόγηση των συνθήκων που θα οδηγούν στην ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού και τους όρους για τη χρηματοπιστωτική βοήθεια να εμπεριέχουν εμπλοκή ανάλογη θεσμικών οργάνων της Ένωσης που θα προσφέρουν έτσι την εμπειρία τους και την προοπτική της Ένωσης. Όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, η παρουσία ενός μηχανισμού υγιού σχετικά με τις τράπεζες περιορίζει το κόστος που έχει σχέση με μια χρεοκοπία τραπεζών στην περίπτωση ενός, ε, μιας ε, διασυνοριακής τραπεζικής ομάδας. Αυτό θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μοιραστεί το δημόσιο κόστος όταν αυτό απαιτηθεί και αν απαιτηθεί. Γι' αυτό είμαστε υπέρ του γενικού πολιτικού στόχου, του νέου πλαισίου για την οικονομική ανάκαψη των τραπεζών και το ψήφισμα που πρότεινε η Κομισιόν. Αν και η εφαρμογή ε, του νέου καθεστώτος ψηφίσματος στην Ένωση ήδη μπορεί να μειώσει το φορολογικό κόστος σε, για χρεοκοπία τραπεζών, πιστεύω ότι θα πρέπει ρητές ρυθμίσεις να υπάρξουν έτσι ώστε στο μέλλον ο χρηματοπιστωτικός ε, κλάδος να φέρει το βάρος ενδεχόμενων νέων κρίσεων. Ως μέρος ενός ε, πλαισίου αξιόπιστου ε, θα είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη και εισφορές των τραπεζών. Αλλά μία εισφορά των τραπεζών θα πρέπει να είναι μόνο ένα συμπληρωματικό εργαλείο σε ένα σύνολο μιας εργαλειοθήκης με στόχο την απορρόφηση των απολειών συστηματικά σημαντικών τραπεζών συγκεκριμένων ε, επιπλέον ε, ε, βάρη στο κεφάλαιο και στη ρευστότητα. Το Financial Stability Board, όπως ξέρετε ήδη, διερευνά διάφορες λύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το μετατρεπταίο κεφάλαιο και διάφορα εργαλεία τα οποία έχουν σχέση με το χρέος. Επικροτώ το ότι η Κομισιόν θεωρεί την εισφορά των τραπεζών bank levies και διάφορα προγράμματα διάσωσης τραπεζών bail-in για, την, για το μελλοντικό πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης στην Ένωση. Η τράπεζα είναι έτοιμη να συμβάλλει στο δύσκολο αυτό έργο, το ακόμα είναι μπροστά μας, όσον αφορά την εξέλιξη αυτού του πλαισίου. Επίσης, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την σημερινή μας συνάντηση ως ευκαιρία για να αναφερθώ και σε άλλο επίκαιρο θέμα, την οριστικοποίηση του προτινόμενου κανονισμού της Ένωσης για τα παράγωγα. Ε, τα central counterparties και τους διάφορους εμπορικούς καταθέτες. Στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής σας για τη σημαντική αυτή νομοθετική πρωτοβουλία θα ξέρουμε ότι λαμβάνονται υπόψη ο σημαντικό ρόλο των κεντρικών τραπεζών προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποδομή των αγορών όσον αφορά τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα. Οι κεντρικέ τράπεζε έχουν αποδείξει το σημαντικό του ρόλο στη χρηματοπιστωτική κρίση και γι' αυτό Πιστεύουμε ότι η συμβολή του στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σωστά αντικατοπτρίζεται στο νέο κανονισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να πάρουν ενεργό μέρος στο νέο πλαίσιο της Ένωσης για του ε, CCP, Central Counterparties, για την έγκριση και την αξιολόγηση κινδύνων των υποδομών, ε, τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών και αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση τρίτων μερών κεντρικών τραπεζών και καταθετών σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών η πρόταση της Κομισιόν για τα colleges προβλέπει κατά την άποψή, μου, την ε, λύση προτιμότερη από τις διμερείς αρχές. Επίσης κύριε Πρόεδρε μου ζητήσετε να πω δύο λόγια για ένα άλλο θέμα τα λεγόμενα ευρωομόλογα. Η Κεντρική Τράπεζα δεν είναι υπέρ της εισαγωγής ευρωομολόγων. Ως εγγυημένα ομόλογα τραπεζών στις σημερινές συνθήκες. Ξέρουμε ότι ο στόχος είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς ομολόγων στην Ευρωζώνη και να υπάρξει και ένας ενδεχόμενος μηχανισμός που θα ελαφρύνει ή θα επιλύει την συνεχόμενη κρίση εθνικού χρέους σε σχέση με την υποστήριξη της αγοράς ομολόγων της Ευρωζώνης. Το κύριο πλεονέκτημα θα είναι να έχουμε περικοπή κόστους μειώνοντας το πριμ ρευστότητα στις αγορές ομολόγων. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί ιδιαίτερα αν τα ευρωμόλογα έχουν καθεστώς benchmark συγκρίσιμο παραδείγματος χάρη με τα αμερικάνικα ομόλογα. Τώρα, όσον αφορά την επίπτωση στι ε, ε, εξελίξει του εθνικού Χρέο, το να περάσουμε στα ευρωομόλογα θα αρθεί η πίεση βραχυπρόθεσμα στι σηματαγορέ, αλλά αν δεν αντικατασταθεί από ένα νέο μηχανισμό, ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μα, θα μειώσει τα κίνητρα για υγιή φορολογική δημοσιονομική πολιτική. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε, η φορολογική δημοσιονομική πειθαρχία κινείται με βάση εσωτερικέ διατάξει μέσω των του θεσμικού πλασίου της διακυβέρνησης, τη συνθήκη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με την αξιολόγηση από τους αποταμιευτές και επενδυτές. Τα κοινά εγγυημένα ομόλογα δεν θα επιτρέψουν στους ε, αποταμιευτές και ε, επενδυτέ να εξολογήσουν τι φορολογικέ πολιτικέ των επιμέρου χωρών. Και επειδή δεν έχουμε πολιτική ομοσπονδία με ομοσπονδιακό ε, προπολογισμό, αυτό ενδεχομένω να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στα κίνητρα και να παρεμποδίσει τα κίνητρα για την δημοσιονομική σόφρονα δράση σε εσωτερικό επίπεδο. Γι' αυτό τα ευρωομόλογα θα είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα αν οι, εθνικές, οι εθνικές φορολογικές αρμοδιότητες σαφώς σε επίπεδο της Ένωσης που θα ήταν ομοσπονδία αλλά ως έχει το θεσμικό πλαίσιο σήμερα πρέπει ακόμα να σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά τη γνώμη μας στη συλλογική διακυβέρνηση και εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών αυτό που θα λέγαμε quantum leap, δηλαδή κβαντικό άλμα, προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση. Ενώσο οι πολιτικές αυτές, επαναλαμβάνω, παραμένουν εθνικές. Αξιότιμες κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περάσουμε αμέσω στις ερωτήσεις. Αξινόμου του στο ΕΡΚ, ο Σόμπορ Γκοζές έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη ερώτηση. Σε δύο τμήματα. Καταρχήν, Αναφέρθηκα σε κάποια μέτρα που προτείνονται για την οικονομική διακυβέρνηση ε, και το σύμφωνο ευρώ. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες επεξηγήσεις και προσθήκες. Και το πιο τεχνικό θέμα είναι η λήψη υπόψη των, χρεών επενδύσεων των κρατών μελών. Μια ερώτηση που σας είχα ήδη υποβάλει, αλλά έχει δημοσία. Αυτό το χρέος, το επενδυτικό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ισορροπιών. Εμείς στο ΕΛΚ σας λέω ξεκάθαρα ότι διστάζουμε κάπως, αλλά θα ήθελα να ξέρω την άποψη του Προέδρου της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. <clears throat> για την ε, διακυβέρνηση. Όπως είπα πριν από λίγα λεπτά, θεωρούμε ότι πρέπει ακόμα να επιτευχθεί πολύ πρόοδος για να αποκομίσουμε όλα τα δάγματα της κρίσης που γνωρίζουμε από το 2007-2008. Λοιπόν, παρόλο που σημειώνουμε κάποιες ε, πρόσφατες πρόοδους, ιδίως όσον αφορά την αντιστροφή του βάρους απόδειξης, το comply or explain έγινε αποδεκτό πια από τις κυβερνήσεις εν μέρει όσον αφορά τη δημοσιονομική υποπτήρια, Παρ' όλα αυτά, σε αυτόν τον τομέα από τις άλλους τομείς, θεωρούμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές δυνατότητες πρόοδου. Και όπως είπα ήδη πλιστάκης, ο τριμερής διάλογος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίω το γεγονό ότι ασκεί την ε, επίδρασή του το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το θέμα των κρατικών επενδύσεων, εγώ θα έλεγα προφανώς θα πρέπει αυτό το χρέος να συμπεριληφθεί φυσιολογικά στην επιτήρηση που κάνουμε. Και είναι σαφές ότι θα τις επομιστούν όλοι οι επενδυτές, ή ε, ε, αποταμιευτές σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να διστάσουμε προφανώς πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη. Είναι χρέη και πρέπει να ληφθούν υπόψη ω χρέη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, second on behalf... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με τον ευχαριστώ. Ο κύριος Σουάνγκογκόγκ. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται τα πνεύματα για μια αύξηση των επιτοκίων λόγω μια αύξηση των τιμών ε, στι ε, πρώτε που μπορεί να έχει επιπτώσει βέβαια στη γενική οικονομία. Αυτό ο πληθωρισμό των τιμών είναι πληθωρισμό κόστους, όχι δημοσιονομικού κόστους όμως. Και γι' αυτό η μόνη θεωρητική μέθοδος που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον πληθωρισμό είναι να ε, προκληθεί αύξηση της ε, ανεργίας πράγμα που θα περιορίσει τους μισθούς και θα μας κάνει να αποφύγουμε το δεύτερο γύρο που πολύ φοβούνται. Ρωτώ λοιπόν εν ώψη της σημερινής οικονομικής πολιτικής και της καταπολέμησης του πληθωρισμού, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί η ενεργεία και να μειωθεί η ανάπτυξη. ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως είπα και εισαγωγικά, σήμερα δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω οτιδήποτε σε αυτά που εξετάστηκαν από το Συμβούλιο των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών που το εξάστησε την περισμένη του συνεδρίαση. Και ξέρετε, στην επόμενη μα συνεδρίαση θα πάρουμε αποφάσει. Αλλά εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που ελέγχθησαν. Είναι ουσιαστικό να κατανοήσουμε ότι σε μια περίοδο όπως αυτή τώρα που υπάρχει σημαντική αύξηση του πληθωρισμού το κύριο πρόβλημα όλων των κεντρικών τραπεζών είναι να αποφυγθούν οι επιπτώσεις δεύτερου χείρου. Δηλαδή να αποφυγθεί εκείνοι που ορίζουν τις τιμές, οι επιχειρήσει δηλαδή που ορίζουν τις τιμές, Επίσης εκείνοι που ορίζουν αυτές τις τιμές, ε, τις τόσο σημαντικές ε, κοινωνικές εταίροι δηλαδή στις διαπραγματεύσεις τους, Όλοι αυτοί θα πρέπει, λέω, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το γεγονός ότι εμείς προσπαθούμε να εγγυηθούμε προς τους πολίτες μία σταθερότητα τιμών. Η σταθερότητα αυτή των τιμών είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ιδίω για τους πιο φτωχού ε, μεταξύ των πολιτών. Τη σταθερότητα των ε, τιμών είναι κάτι που παρακολουθούμε πολύ στενά για τους πολίτες μας αυτούς. Και στο παρελθόν καταφέραμε, επίσης σε δύσκολες περιόδους, να διατηρήσουμε τη σταθερότητα αυτή των τιμών και να αποφύγουμε τις επιπτώσεις του δεύτερου γύρου. Ξέρετε ότι τα 12 πρώτα χρόνια του ευρώ είχαμε μέσο όρο πληθωρισμού ετησίως 1,97% και 97% στο τέλειο του περασμένου όρου, κάτω από το 2% δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην υπάρχουν επιπτώσεις δευτέρου γύρου σε αυτή τώρα την τρέχουσα περίοδο που αντικειμενικά είναι μια πολύ απαιτητική χρονική περίοδο. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Εξεπλέχει λίγο με την αιτιολόγηση που δώσατε κατά των ευρωομολόγων. Ξέρω βέβαια τις συζητήσει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Μπορώ να καταλάβω ότι θα πρέπει να είμαστε συνετοί, ιδίω σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένε χώρε ε, τη ζώνη ευρώ έχουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα και έχω κάθε σεβασμό το σημαντικό συνταγματικό δικαστήριο τη Γερμανία. Αλλά αναρωτιέμαι θα είχαμε ε, προχωρήσει στο ευρώ τότε, είχαμε πει ότι θα περιμέναμε να υπάρχει μία ε, συναγματική ομοσπονδιακή ένωση πρώτα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν τρόποι δημιουργίας αυτών των μέσων με πλεονεκτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εγώ σέβομαι εκείνους που από πριν, ε, πριν από 20 χρόνια ήταν τολμηροί και έκαναν κάτι που τότε δεν φαινόταν και πολύ εφικτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Εγώ σας έδωσα την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη τι είδαμε στο παρελθόν, ότι η κρίση δηλαδή προχώρησε με μεγάλη ισχύ όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλες τις ε, ανεπτυγμένες χώρες γιατί όλες οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς όλες έχουν σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα και ξέρετε ότι η παγιωμένη ζώνη ευρώ αντιμετωπίζει μια κατάσταση πολύ καλύτερη σε αυτή την κατεύθυνση από εκείνη στη ΣΥΠΑ. Και σύμφωνα με τις σημερινέ προβλέψεις θα υπάρχει ένα ετήσιο έλλειμμα της ε, ζώνης ευρώ που θα είναι περίπου το ίμιση από κοινό των ΙΠΑ ή της Ιαπωνία. Είναι λοιπόν ένα κεντρικό, κεντρικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα ε, ίδρυσης της ε, Ευρώπης, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και γενικά των ανεκτημένων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τις χώρες αυτές προς την καλή κατεύθυνση. Και εκεί που νομίζω συμφωνούμε και για την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης και όσον αφορά τον προϋπολογισμό και όσον αφορά την επιτήρηση των μακροοικονομικών πολιτικών, είναι σαφές ότι εμείς στο Συμβούλιο δικητών Τραπεζών θεωρούμε ότι ακριβώς θα παίξει, να, πρέπει να παίξουν ένα ρόλο και οι αποταμιευτές και οι επενδυτές για να πιέσουν ορισμένες χώρες, όλες τις χώρες ε, και τα κοινοβούλια τους προς την οδό της σοφίας. Καταλαβαίνω λοιπόν τις ε, προτάσεις που έγιναν από ορισμένους, αλλά δεν είναι αυτή η δική μας θέση να σας ευχαριστώ. Την Ισιάρη Βίκη. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας κύριε Τρισέ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχετε να πείτε πάντα. Εγώ εκπροσωπώ 9 ε, χώρε στην ομάδα μου, εκ των οποίων οι 7 δεν χρησιμοποιούν το ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ. Και εγώ συγγήτρια για τα δημοσιονομικά έχω ήδη υποβάλει τι τροπολογίε που ζητήσατε ανεξάρτητα τούτο για ε, εποπτεία που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στις ε, χώρες Λοιπόν, πραγματικά παρακολουθούμε ακριβώ τι γίνεται. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που μα ενδιαφέρει όλου: το θέμα των τραπεζών και των τραπεζών που εργάζονται δυσυνοριακά. Ορισμένοι από εμά εξεπλάγημεν ότι δεν υπήρχαν περισσότερα για ομόλογα στην προηγούμενη, την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση των χωρών ευρώ. Θέλω να μας πείτε κάτι παραπάνω. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα ότι υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι για τις ε, πτωχεύσεις. Ε, ε, δεν υπάρχουν παντού μαχανισμοί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας ε, των τραπεζών. Αυτό όμως κατά τη γνώμη μου θα ήταν ουσιαστικότατο για να φροντίσουμε ο φορολογούμενος να μην είναι εκείνο που πάντα θα πρέπει να επομισθεί αυτό το άκτο. Συμφωνείτε? Απάντηση. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ομολογώ ότι συμφωνώ απόλυτα ότι και στο επίπεδο της Ευρώπης και παγκόσμιος, θα ήταν σημαντικό να έχουμε στον κατάλληλο συντονισμό των κανόνων πτώχευσης για Ινστιτούτα που εργάζονται ε, διασυνοριακά, όπως είπαμε. Είδαμε τι έγινε μετά τις τραγικές ε, εξελίξεις ε, μέσω Σεπτεμβρίου του 2008. Τα προβλήματα δεν είναι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο και σε σχέση με την Επιτροπή Βασιλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι σαφές ότι εφόσον έχουμε ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία και έχουμε διασυνοριακά δημοσιονομικά Ινστιτούτα και χρηματοπιστωτικά Ινστιτούτα είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό, Ευρωπαϊκό και διεθνώ. Δεν είναι εύκολο, αλλά υποστηρίζει απόλυτα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι προσπάθειε για πρόοδο προ την κατεύθυνση αυτή, που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Εάν στο μέλλον θέλουμε να αποφύγουμε νέες τεράστιε δυσκολίες, όπως εκείνε που είδαμε στο παρελθόν και ιδίω όταν επιτόχευσε η Lehman Brothers γιατί ήταν σαφές ότι οι κανόνες από την άλλη όχθη του Ατλαντικού ήταν πολύ διαφορετικοί από τους δικούς μας κανόνες εδώ. Οι διαφορές μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου ήταν τεράστιες. Λοιπόν δεν είναι ευρωπαϊκό αλλά παγκόσμιο το πρόβλημα αυτό. Ιδίως για τις προηγμένες οικονομίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξενόμενος τον πολύ. Φιλίπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπατε για τα ουσιώδη δυστυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ότι υπάρχει ένα ε, δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το ίμιση καλύτερο από τον ΙΠΑ και της Ιαπωνίας, αλλά όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο υπάρχει επίσης μια ισορροπημένη κατάσταση. Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, επανέλθουν στην ανταγωνιστικότητα ορισμένε χώρε που δεν είναι ανταγωνιστικέ αυτέ. Υποθέτω ότι εννοείται θα πρέπει να εξάγουν. Ε, αυτό σημαίνει όμω ότι θα πρέπει να εξάγουμε προ τα έξω, γιατί δεν οφείλει να εξάγει ο ένα προ τον άλλον. Δηλαδή, ε, προσπίζεται μια Ευρώπη που θα έχει ένα γενικό εμπορικό πλεόνασμα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια διαφορά μακροοικονομική, δηλαδή υπάρχει ε, ανάπτυξη στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες, ακόμα έφεση σε άλλες χώρες. Τι πιστεύετε θα πρέπει να γίνει για να υπάρχει καλύτερος πολιτικός ε, ε ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι οικονομίες της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Βελγίου κλπ. Απάντηση. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Έχω να πω και αυτό δεν είναι μόνο η θέση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και όλων των κυβερνήσεων. Και όπω είπατε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ότι να ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων και έτσι να επιτραπεί στου Ευρωπαίου να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη απασχόληση, ε, ψηλότερο επίπεδο ζωής κατά κεφαλή και να βρεθούν σε καλύτερη κατάσταση παραμένω σε κάποια ισορροπία. Θεωρώ λοιπόν ότι η αύξηση της αναγνωσικότητας, η βελτίωση της αναγνωσικότητας είναι πραγματικά μία δυνατότητα για να βελτιωθεί η απασχόληση και το επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων. Είναι σημαντικό αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας. Και έτσι ε, νομίζω ότι βελτιώντα την αγωνιστικότητα μας θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να αυξήσουμε την απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά είναι σημαντικό ότι πρέπει να είμαστε σε μια ισορροπία και θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι της Δένης Ευρώ θα παραμείνουν σε ισορροπία γιατί αυτό είναι λίγο πολύ σύμφωνο με την ιστορική του στάση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συλλογικά δεν βρισκόμαστε σε μεγάλη ανισορροπία. Σχεδόν σε ισορροπία βρισκόμαστε μόνιμα. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι με μια στρατηγική μακροπρόθεσμη ε, πολιτική. πολιτικής θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα πλεόνασμα παρά το αντίθετο στις τρέχουσες πληρωμές γιατί βλέπουμε τις ε, αναπτυγμένες χώρες που έχουν μόνιμα εξωτερικά ελλείμματα. Δεν είναι αυτό ίσως καλό. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις συντάξεις σε, μια πυραμίδα ηλικίας ε, τα επόμενα έτη. Στον αφορά τη δεύτερη σας ερώτηση, θα έλεγα στα σύντομα ότι στην ζώνη ευρώ βρισκόμαστε σε μια ζώνη στην οποία η νομισματική πολιτική είναι ένα δεδομένο και είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ ενώπιον ημών να επαναλάβω το γεγονό ότι μπορέσαμε να δώσουμε για 12 χρόνια στον Ευρωπαίο πολίτη τη σταθερότητα τιμών που ήθελε και που ήταν ευθυγραμμισμένο με αυτό που είχε παρατηρηθεί σε πολλέ χώρε, δηλαδή κάτω το 2%, σχεδόν 2% πληθωρισμό. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ε, βέβαια καταστάσεις ε, στις οποίες τα άλλα μέσα της οικονομικής πολιτικής που διαθέτουν οι κυβερνήσεις να χρησιμοποιηθούν όσο δυνατόν πιο ενεργά. Δημοσιονομική πολιτική, διαστρατική πολιτική, τα μηνύματα που μπορούν να προσταλούν να αφορά την ανάπτυξη του κόστου σε μια οικονομία. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στα μέτρα που μπορούν να υιοθετηθούν όσον αφορά τους ε, κανόνες ε, της ασφάλισης, ε, γιατί είδαμε ότι συστηματικά οι κανόνε αυτοί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Αν δεν του έπαιξαν στο παρελθόν θα πρέπει να του παίξουν στο μέλλον. Thank you very much. I've got the GUI next. Ευχαριστώ. Ο Μιγγέλ Πόρτα ε, λέει εδώ από την Ενωτική Αριστερά, δεν τον βλέπω. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που ε, είστε ε, εδώ παρόν κύριε Τρισέ για τη συζήτηση. Κύριε Τρισέ, τονίζετε πάντα την αξιοπιστία του δημοσίου, δεν χωρά καμία αφιβολία ότι είναι χρήσιμη και σημαντική. Το είχα πει και στο παρελθόν. Το πρόβλημα όμως της υπερβολικής χρέωσης ή το σημερινό υπερβολικό χρέος οφείλεται κυρίως σε μια κρίση των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού στήματος και όχι κρίση αξιοπιστίας ε, του κράτους. Το moral hazard είναι ένα θέμα τραπεζών, όχι κρατών. Εκεί τίθεται το πρόβλημα στην αξιοπιστία των τραπεζών. Και θα πρέπει να τονιστεί πολύ περισσότερο και με πιο σαφέστερο τρόπο ότι πρόκειται για την αξιοπιστία των τραπεζών το κράτος στάθηκε αξιόπιστος εταίρος και παραστάσεις στο πλευρό των τραπεζών όταν το χρειάστηκαν. Και θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση με ένα μικρό σχόλιο για τα ευρωομόλογα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ε, από τη δική σας σκοπιά, αλλά δεν θα ήταν πολύ πιο μεγάλη βοήθεια και πιο σημαντική ε, με τα ευρωομόλογα να βοηθήσουμε τις υπερχρεωμένες χώρες για να αποπληρώσουν το χρέος. Την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν τα όσα οφείλουν τα κράτη αυτά με τα ευρωομόλογα. Θα τους βοηθούσαν πολύ περισσότερο από ό,τι αυτό κάνουμε τώρα. Και για την Ιαπωνία, το είπατε και στην αρχή. Τώρα οι ανάγκες ε, οι πιστοτικές της ε, Ιαπωνίας ε, μπορεί να οδηγήσουν στα ύψη τα επιτόκια. Αυτό το έχετε σκεφτεί. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση στα αγγλικά. Αυτό που μόλις είπατε για το χρηματοπιστωτικό τομέα τα προσυπογράφω. Έδειξε μία ευαισθησία και ένα επίπεδο πώς να το πω, ένα τόσο εύθραυστο χαρακτήρα που δεν επιτρέπεται και κάλεσε όλα τα κράτη ε, των προηγμένων οικονομιών ας πούμε να βοηθήσουν για να μην έχουμε τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κρίση από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξάγουμε όλα τα διδάγματα ε, από τα όσα συνέβησαν. Τούτο λεχθέντον όμως ισχύει και κάτι άλλο για όλες τις προηγμένες οικονομίες. Όταν αρχίζει κανείς να εξετάζει την κατάσταση αναχώρα, υπάρχουν χώρες που έχουν προβλήματα και αυτό μπορεί να είναι αποκλειστικά λόγω ε, της κρίσης των τραπεζών, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που ε, ακολουθούν κακή, ε, δημοσιονομική πολιτική. Γι' αυτό έχουν προβλήματα και αυτό ισχύει και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και επίσης ε, αναγνωρίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και προς τις δύο ε, κατευθύνσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο που επιμένετε και στην τραπεζική διάσταση και νομίζω ότι θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί και να φροντίσουμε και τη δημοσιονομική πολιτική. Ε, εν πάση περιπτώσει αποφύγαμε μια τρομακτική ε, καταστροφή που θα μπορούσε να επέλθει διότι οι υπογραφές των κρατών ήταν αξιόπιστες σε περιόδους κρίσης. Εάν δεν είχαν τα κράτη τότε πρόσωπο, τότε θα ήμασταν πραγματικά σε μια πάρα πολύ δινή κατάσταση, σε μια τρομακτική καταστροφή. Δηλαδή, ακριβώς επειδή στο μέλλον δεν αποκλείεται τίποτα, θα ε, εξάγουμε όλα τα σωστά και τα απαραίτητα διδάγματα από την κρίση αυτή και θα πρέπει η υπογραφή ε, κάθε κράτους να είναι εγγυητής και αξιόπιστη, όχι μόνο της Ευρώπης και μιλώ για όλα τα κράτη του κόσμου, για να ε, υπερβούμε οποιαδήποτε πιθανή δυσκολία στο μέλλον. Για τα ευρωομόλογα, για το σχόλιο που κάνατε, εξήγησα προηγουμένως γιατί θεωρούμε εμείς ότι επί του παρόντος δεν είναι ε, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε. Κατανοώ το επιχείρημά σας, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε πεπισμένοι ακόμα. Και σαθμίζουμε αναλόγως ε, όλα τα επιχειρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει κύριος Μπάλτς. Έχω δύο ερωτήσεις, μία για την Ιαπωνία. Ε, στις πιο πρόσφατες ε, παρεμβάσεις ακούσαμε ότι θα πρέπει να μειωθεί το γεν που είναι πολύ υπερτιμημένο για να βοηθηθεί και η οικονομία. Την Παρασκευή όμως η Κεντρική Τράπεζα ε, έστειλε δισεκατομμύρια γεν για να τονώσει το σύστημα και να αποφύγει η κατάρρευσή του. Εσείς Πώς το εκτιμάτε αυτά. Ε, είναι πάλι το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα υποπίεση μετά από τις εξελίξεις αυτές. Και μετά ε, η οικονομία είχε αρχίσει σιγά σιγά να ανακάμπτει από την κρίση. Τώρα με τα γεγονότα στην Ιαπωνία ε, δεν θα επηρεαστεί και μάλιστα πολύ ουσιαστικά. Έχω και άλλη μια ερώτηση. Η θητεία σας κύριε Πρόεδρε δυστυχώς λύγει τον Οκτώβριο. Νομίζω και μερικοί άλλοι συνάδελφοι έχουν την ίδια άποψη με μένα. Και επειδή είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς προσωπικά τώρα, ποιες προτεραιότητες έχετε για τους υπόλοιπους μήνες που σας μένουν, έτσι ώστε να παραδώσετε στο διάδοχό σας όχι απλώς μια ε, καλώς διοικούμενη τράπεζα που σίγουρα θα το πράξετε, αλλά και να είναι και προετοιμασμένη για να περάσει το δύσκολο χειμώνα που επίκειται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την Ιαπωνία πρώτα. Όπως είδατε την περασμένη εβδομάδα, επετέχθη συνένεση μεταξύ ε, της εκτελεστικής εξουσίας και ε, των διοικητών των κεντρικών τραπεζών του ε, G7 για να συμφωνήσουμε και να στείλουμε το σωστό μήνυμα στις αγορές. Στο εσωτερικό των ε, βασικότερων συναλλαγμάτων και νομισμάτων. Ήταν ο σωστός τρόπος, θεωρήσαμε, για να αντιδράσουμε ε, με βάση τις εξελίξεις. Εγώ δεν θα ήθελα να επεκταθώ ως προς τον αντίκτυπο των τεκτενομένων ε, στην ίδια την Ιαπωνία. Βεβαίω προσεκτικά, πολύ προσεκτικά παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν και τι αντίκτυπο έχουν στην Ιαπωνική οικονομία και ενδεχομένω σε κάποιους εταίρους της Ιαπωνίας. Είχαμε το προηγούμενο του Κομπέ και τώρα θα πρέπει να δούμε σε ποιο τομέα, ας πούμε, σε ποιο βαθμό ε, είναι διαφορετική η κατάσταση. Είναι γεγονό ότι η ανθρώπινη τραγωδία είναι ανίποτη. Η συνήθις κατάσταση μετά από μια τέτοια τραγωδία ποια είναι. Στην αρχή υπάρχει μεγάλη πτώση της δραστηριότητας που συνδέεται άμεσα με τις δραματικές αυτές εξέλιξεις, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αυτή ε, απορροφάται και αρχίζει η ανάκαμψη, η ανοικοδόμηση που από την ίδια της τη φύση αναθερμαίνει τις δραστηριότητες οικονομικές. Ε, είναι πολύ ευαίσθητη η ισορροπία να εκτιμήσει κανείς σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, αλλά το μελετούμε και το παρακολουθούμε από πολύ κοντά και επιπλέον έχουμε και το πυρηνικό ζήτημα που δεν είναι μόνο η ιαπωνική υπόθεση αλλά και παγκόσμια και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αναθερμανθεί παντού και συζητείται. Για τη δεύτερη ερώτησή σας ήθελα να σας πω το εξής. Με ρωτούν από καιρούς καιρών η παρούσα περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική κτλ ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι όλοι οι καιροί είναι απαιτητικοί. Από τότε που εισήχθη το ευρώ μέχρι που έσκασε η φούσκα.com μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου ε, ε, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις πάρα πολύ δύσκολες ε, σοκ πετρελαϊκό εμπορευμάτων και επίσης δεν σας κρύβουμε ότι η κρίση του 2007 και του 2008 είναι πάρα πολύ απαιτητική και γενικά η καιρή είναι απαιτητική όλο το διάστημα. Εγώ τη δουλειά μου θα συνεχίσω να κάνω μαζί με όλους τους συναδέλφους. Όπως γνωρίζετε όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε από τους έξι ε, του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από τα ε, μέλη ε, του Ευρύτερου Συμβουλίου που είμαστε 23. Είναι δύσκολη η περίοδος, ε, θα αναλάβουμε τις ευθύνε μας όπως πράττουμε πάντα. Άλλωστε αυτό ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα. Για όλα τα θεσμικά όργανα είναι κερία απαιτητική. Και επίση ε, με ρωτήσατε, να επικεντρωθώ σε ένα σημείο, σε τι θα μπορούσα να θέσω ως προτεραιότητα. Αν ε, θα μπορούσε να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη βελτίωση την οποία και εσείς συζητάτε στη ε, οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης και των 27 και των 17 σημαίνει ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας και για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, για το απότερο μέλλον. Ο Έντουαρτ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Μια σύντομη ερώτηση. Κύριε Τρισέ, η Κεντρική Τράπεζα είναι ευχαριστημένη με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χειρίζονται τα θέματα αφαιρέγγιων τραπεζών όπως η Anglo-Irish Bank. Έχετε καμία σύσταση για το μέλλον, αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Τρίσε. Για το μέλλον, πρόθεσμα εργαζόμαστε για το θέμα αυτό συνολικά όπως σας είπα με το μηχανισμό FSB και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να έχουμε συντονισμένες έννοιες που θα ισχύουν για όλους συνολικά και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και φυσικά για την Ευρώπη. Όσον αφορά την άμεση απάντηση εκ μέρου τη Ιρλανδική κυβέρνηση σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Κομισιόν και την Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχω κάποιο ειδικό σχόλιο να κάνω. Ο Ρέμο για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, η Ισπανία παραμένει στην οικονομική κρίση τους δύο πρώτους χρόνους φέτος δεν αυξάνονται οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις, ο δείκτης ανεργίας ανεβαίνει, παρά το ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στην Ισπανία από πέρυσι. Πρώτη ερώτηση, υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απόκλησης στην Ευρωζώνη. Δεύτερη ερώτηση, στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα ανεβάσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες, τι επίπτωση θα έχει αυτό στην Ισπανική οικονομία. Και τρίτο, οι ισπανικές περιφέρειες φέτος θα χρειάζονται περίπου 21 δις ευρώ για φέτος. Η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί το ενδεχόμενο να διασώσει μερικές ισπανικές περιφέρειες στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Πρώτη παρατήρηση. συχνά με ρωτάνε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας που έχετε ένα νόμισμα. Έχετε τη Γερμανία που ε, ε, πάει προς τα πάνω και την Ισπανία και μερικές άλλες χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση όπου η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτική. Με ρωτάνε. Και απαντώ Είχα ακριβώ το αντίστροφο ερώτημα πριν. Πώς είναι δυνατόν, μου λέτε, να διοικείται μια χώρα με ένα νομισμό όπου η Γερμανία είναι τραγικά επίπεδο και η Ισπανία έχει μια, ένα δίκτυ πολύ προ τα πάνω. Ε, λοιπόν, όταν έχουμε τεράστιες οικονομίες, 300 εκατομμύρια άνθρωποι, 350 εκατομμύρια στην περίπτωσή μας, μιλάω για Αμερική και Ευρώπη, υπάρχουν χώρες που για διάφορους λόγους η κάθε μία βρίσκονται στη διαφορετική κατάσταση. Η μία σε σχέση με την άλλη η Ισπανία και η Γερμανία πάνω κάτω είναι στην αντίστροφη κατάσταση σήμερα σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια. Είναι ακριβώς η ίδια διακύμανση. Αυτή βλέπουμε και, τη μεριά, και στη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας το αναφέρω εμπαρόδο ότι εξορισμού βρισκόμαστε σε μια πολύ ευρεία οικονομία και χαίρομαι για το ότι η Γερμανία δούλεψε, ξανακέρδισε την ανταγωνιστικότητά της και τώρα έχει την οικονομική εξέλιξη που έχει, την οικονομική ανάπτυξη που έχει. Αυτό είναι καλό και για την Ισπανία. Ήταν καλό για την Ισπανία όταν η Ισπανία είχε γρήγορη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έμεσα βοηθούσε όλη την Ευρωζώνη. Βέβαια, τούτων δεδομένων η Ισπανία πήρε μερικές σημαντικές αποφάσεις για βελτίωση και αυτές οι αποφάσεις και οι δρόμοι που διάλεξε δεν είναι εύκολοι δεν, δεν θα δώσουν άμεσα αποτελέσματα αλλά κινούνται στη σωστή κατεύθυνση Τώρα, για την νομισματική μας πολιτική είπα, δεν έχω να προσθέσω τίποτε σε αυτά που είπα στις αρχές Μαρτίου. Επαναλαμβάνω μόνο ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε σταθερότητα τιμών για όλη την Ευρωζώνη. Το 1,97% που ανάφερα ήταν για όλη την Ευρωζώνη. Και επιβάλλεται να το πετύχουμε αυτό γιατί αυτό μας ζητάνε οι συμπολίτε μας. Και γιατί το λένε οι συνθήκες και γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους τους συμπολίτε μας, ιδιαίτερα για τους πιο φτωχούς και τους πιο τροτούς και ευάλωτους. Γι' αυτό οι αποφάσεις μας έχουν πάντα σαν γνώμονα τη σταθερότητα των τιμών που με τη σειρά της έχει σημαντική επίπτωση γιατί όπως ξέρετε όλα τα επιτόκια όλη της Ευρώπης στηρίζονται στην προσθήκη στους, στα πραγματικά, στους πραγματικούς συντελεστές πληθωριστικές προσδοκίες τα επόμενα χρόνια και στο πριν κινδύνου. Αν πάρουμε λοιπόν τις πληθωριστικές προσδοκίες και αν αυτές αυξάνονται, άμεσα τα επιτόκια μέσω μακροπρόθεσμα αυξάνονται και αυτά. Συγγνώμη, τα βράχη μέσω πρόθεσμα αυξάνονται και αυτά. Και δεν το θέλουμε αυτό, τουλάχιστον στις σημερινές συνθήκες. Γι' αυτό επιβάλλεται να παραμείνουμε στην άγκυρα αυτή που έχουμε σταθερές επιθεωριστικές προσδοκίες. Τώρα για το bailout, για την διάσωση που είπατε, δεν έχω να κάνω καμία σύσταση για την Ισπανία. Με ρωτήσατε για τις περιφερειές, για τις περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές, περιφερειακές. Φυσικά όχι. Φυσικά δεν προβλέπουμε σε καμιά περίπτωση να εμπλακούμε σε τέτοιου είδους δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για το ομάδα ECR, ο Ντέρκ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αν εγκρίνει τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας τότε το Ταμείο Διάσωσης τη Ευρωζώνης θα μπορεί να παρέμβει στην πρωτογενή αγορά. Η συμφωνία όμως δεν δίνει το δικαίωμα αγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Τη λύση αυτή ξέρουμε ότι είναι υποστήριξη και δική τράπεζα. Ένα άλλο εργαλείο που λείπει είναι η δυνατότητα να επεκταθούν βραχυπρόθεσμα δάνεια σε χώρε που προσωρινά χάνουν την πρόσβαση στη ρευστότητα. Κύριε Πρόεδρε, Ποια είναι η γνώμη σας για το εύρος του Ταμείου Διάσωσης της Ευρωζώνης όπως προβλέπετε στην μέχρι τώρα πρώτη συμφωνία. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα θυμόσαστε η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ήταν το Ταμείο αυτό και το σημερινό και το μελλοντικό να βελτιωθεί και ποσοτικά και ποιοτικά. Ποσοτικά αυτό που αποφασίστηκε από την εκτελεστική εξουσία κατά τη γνώμη μας είναι στο ύψος αυτού που είχαμε κατά νου. Και όσον αφορά το Ταμείο Σταθεροποίησης, το σημερινό και το μελλοντικό, τα 500 δις κατά τη γνώμη μας, είναι στο ύψος της ε, φερεγγιότητας και δεν διστάζω να το δηλώσω αυτό. Όσον αφορά την ευελιξία, υπάρχουν στοιχεία βαθμοί ευελιξίας που εισήχθησαν στην απόφαση καταρχή και άλλα στοιχεία ευελιξίας που τα αναφέρατε κι εσείς, παραδείγματο χάρη η παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά. Αυτά δεν ε, είναι σύμφωνα με αυτό που εμείς ε, προτείναμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Γιατί όλα αυτά είναι δημόσιες δηλώσεις μου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Πρόεδρος για το ΕΛΚ, Χωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και χίλια συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση. Η καθυστέρηση στο αεροπλάνο. Δεν έφταιγα εγώ. Για το μόνιμο μηχανισμό διάσωσης έχω μια ερώτηση. Η καγκελάριος Μέρκελ το Νοέμβριο δήλωσε στο G20 ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα κληθούν να υποστηρίξουν τμήμα του κόστους για τη διάσωση. Μα ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας νόμιζα ότι είχε πει ότι αυτό θα σήμαινε πολύ μεγάλη αστάθεια, απτητικότητα των αγορών και θα εκτόξευε στα ύψη τα επιτόκια. Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι θα γινόταν απερίπτωση από το 2013 και μετά και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η μόνη περίπτωση που γνωρίζω εγώ αντίστοιχη ήταν ε, η Αργεντινή το 2004 που παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα το ζήτημα, δεν λύθηκε. Πώς βελτιώνει λοιπόν αυτό την κατάσταση, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα να συμμετέχουν στο μόνιμο πλέον μηχανισμό διάσωσης και ιδιώτες. I uh, Απάντηση. Έχω, υπήρξε ένα κείμενο που εγκρίθηκε από ό,τι ξέρω από όλες τις κυβερνήσεις, τις ενδιαφερόμενες, 28 Νοεμβρίου πέρσι, όπου σαφώς δηλώνεται ότι οι Ευρωπαίοι θα ακολουθήσουν τους ε, καθολικούς κανόνες του ΔΝΤΑΦ όσον αφορά το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Και δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Εξάλλου, ε, οι, οι Πρωθυπουργοί επανέλαβαν τη δήλωση αυτή στην πρόσφατη συνάντησή τους και μάλιστα δημοσίευσαν ως παράρτημα στο, στην ανακοίνωσή τους αυτό τον κώδικα που κατά τη γνώμη μου, εξορισμού βέβαια, είναι η θέση των Ευρωπαίων. Επιβεβαιώθηκε και πάλι ε, επίσημα, επανελήφθη η δήλωση. Και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε ότι αυτό ήταν μια χρήσιμη διευκρίνηση, διότι μας λέει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν τους ίδιους κανόνες με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. για αυτούς που βάζουν αυτή, όπως σας είπα, την εθνική υπογραφή σε παγκόσμιο επίπεδο για την ομάδα ε, των ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών Γκουάμ. Κύριε Πρόεδρε, η Βρετανική και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα είναι αρκετά ε, καλυμμένη, μπορούν να περάσουν άνετα το χειμώνα γιατί μπορούν να χρηματοδοτήσουν με το δικό τους νόμισμα το δημόσιο τους έλλειμμα, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Ενώ το καθεστώς της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το απαγορεύει αυτό. Ωστόσο, στη δευτερογενή αγορά αγόρασε εθνικό χρέος η Κεντρική Τράπεζα πριν από μερικές εβδομάδες. Η Κεντρική Τράπεζα σταμάτησε να αγοράζει το ελληνικό εθνικό χρέος και τα επιτόκια για τα διετή δάνεια της Ελλάδας αμέσως πήδησαν στο 15%. Κατά τη γνώμη σας υπάρχει σχέση αιτιολογική, αιτιώδης μάλλον μεταξύ των δύο ή η μακροοικονομική κατάσταση Ελλάδας ήταν τέτοια που θα έπρεπε μέσω πρόθεσμα να προβλεφθεί μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Απάντηση. Όπως ξέρετε έχουμε ένα δόγμα στην Κεντρική Τράπεζα που λέει διαχωρίζουμε όσο πιο αυστηρά γίνεται τα μέτρα νομισματικής πολιτικής, τα λεγόμενα στάνταρ, επιτόκια δηλαδή, που καθορίζονται προκειμένου να έχουμε σταθερότητα τιμών, μέσω πρόθεσμα όπως ορίζει η συνθήκη, και αυτό μας ζητάνε και οι συμπολίτε μας, και απ' την άλλη έχουμε τα λεγόμενα μη στάνταρ μέτρα, τα οποία εισήχθησαν από τότε που χτύπησε στις αγορές η κρίση και που οδήγησαν σε ορισμένες αγορές ε, να υπάρξουν συμπεριφορές ανώμαλες, πολύ ανώμαλες. Μεταξύ αυτών των μέτρων, των μη στάνταρ, non στάνταρ, είναι παραδείγματο χάρη η εκχώρηση ανεφόρου ρευστότητας, full allotment, σε σταθερή τιμή, είχαμε τότε επαναχρηματοδοτούμε για έξι μήνες ένα χρόνο τις τράπεζες, τώρα αυτό σταμάτησε. Είχαμε παρεμβάσει στην αγορά των coven bonds, των ομολόγων, και είχαμε και ένα πρόγραμμα που το λέμε SMP, στο οποίο εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε. Όλα αυτά τα μέτρα, τα μη στάνταρ, σε κάθε περίπτωση έχουν σαν στόχο να έχουμε μια καλύτερη εφαρμογή της νομισματικής μας πολιτικής. Οι συνθήκες παραμένουν περίπλοκες όσον αφορά τη λειτουργία των αγορών. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου, όπως σας είπα στην εισαγωγή μου, κρατήσαμε για το επόμενο τρίμηνο τα μη πρότυπα μέτρα παροχής ρευτότητας σε τρεις μήνες με βάση το full allotment όπως σας είπα αυτά τα μέτρα έχουν σε στόχο να μας επιτρέψουν να αποκαταστήσουμε όσο γίνεται δεδομένων των ανώμαλων συνθήκων κατά τις οποίες κινούμαστε τους διάβλους διαβίβασης και εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και πάλι για το ΕΛΚ η Ρόδη Κράτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είχα σκοπό να ρωτήσω για τα ευρωομόλογα, αλλά δώσατε σαφείς ε, απαντήσεις, όπως και για τον μηχανισμό στήριξης ε, της σχέσης του με την αγορά ε, ομολόγων κρατών από την ανοιχτή αγορά. Οπότε θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, το σύμφωνο για το ευρώ. Πιστεύετε ότι όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα ε, θα δώσει μια προστιθεμένη αξία στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης ε, το οποίο ήδη είναι σε επεξεργασία και ελπίζουμε γρήγορα να καταλήξει σε μια συμφωνία. Και δεύτερον, η διαφαινόμενη αύξηση των επιτοκίων. Έχετε, ε, υπάρχουν μελέτες ότι δεν θα επιβαρύνουν την ανάκαμψη της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το, για το πρώτο σημείο βέβαια θα πω ότι υπάρχει μια πρόοδος και θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί η πρόοδος γενικά, ακόμα και πρόσφατα όσον αφορά την ποιότητα της διακυβέρνησης των 27 και των 17. Το τελευταίο. είναι μια ενεξελίξη πρόοδος και βέβαια σχολείται το Κοινοβούλιο με τη συζήτηση αυτή για την διακυβέρνηση και θα έλεγα ότι πραγματικά βασιζόμαστε πάρα πολύ στην εργασία σας και στη συνεργασία σας επίσης με τα άλλα θεσμικά όργανα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για το δεύτερο σημείο θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι εμείς καλούμεθα να προσφέρουμε ε, σταθερότητα τιμών σε 531 εκατομμύρια πολιτών. Πολύ σημαντικό το κάναμε στο παρελθόν, το ξανακάνουμε στο μέλλον. Και αυτό είναι μια προϋποθέτηση για α, βιώσιμες θέσεις εργασίας και δημιουργία απασχόλησης στο μέλλον. Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα δείτε ότι το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον του ευρωχώρου θα καταρρεύσει. Γιατί ακριβώς οι ε, προσδοκίες πληθωρισμού θα είναι υψηλότερες. Γι' αυτό η σταθερότητα αυτή των τιμών ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και σχετίζεται και με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εμείς ε, πληρούμε έτσι ένα από τους όρους για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Πάλι οι σοσιαλιστές. Κύριε Τρισέ, ε, αυτή τη στιγμή έχουμε χώρες χρεωμένες που απειλούν την σταθερότητα του ευρώ και προσπαθούν να μην χρησιμοποιήσουν το προσωρινό ταμείο σταθερότητας. Αν ανιστρέπταμε τα πράγματα, τι θα γινόταν και εξετάσουμε το μόνιμο μηχανισμό σταθερότητα. Και έχουμε μια κατάσταση στην οποία ορισμένε χώρε βρίσκονται σε κρίση και χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν αυτό το ταμείο χωρίς να απειλούν τη σταθερότητα του ευρώ, επειδή είναι πολύ μικρές χώρες. Θα πρέπει νομίζω να ωφεληθούν από το ταμείο αυτό, έχοντα συμβάλει προ αυτό βέβαια. Απάντηση. Καταρχήν, θα ήθελα να πω, αυτή είναι μια απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί από τους αρμοδίους. Εμείς δεν είμαστε τμήμα της λήψης απόφασης αυτής. Πρώτον αυτό. Δεύτερο. Ο Λούκληρη Ευρώπη βασίζεται στην ιδέα ότι όλες οι χώρες βρίσκονται επί ίσης όρης και τη χανοτσίδης μεταχείρισης άσχετα με το μέγεθός τους. Αυτό ισχύει για όλους τους κανόνες διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των μικρών και των μεγάλων και των πολύ μικρών χωρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι μπορεί μια χώρα να είναι μικρή και παρ' αυτά να είναι ορατή και να δημιουργεί προβλήματα. Όχι για το ευρώ ίσως, αλλά για την ε, οικονομική σταθερότητα του συνόλου του ευρωχώρου. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση αυτή μεταξύ του ευρώ αυτού καθεαυτού ένα νόμισμα που βασίζεται στο γεγονός ότι, όπως σας είπα, εδώ και 12 χρόνια μπόρεσε να διατηρήσει ένα εντυπωσιακό επίπεδο σταθερότητας τιμών, καλύτερο από εκείνο που είχαμε τα 50 χρόνια πριν από αυτό. Και θα μπορούσα να φανταστώ επίσης ότι η Ευρώπη στο σύνολό της και όσον αφορά τους τρέχοντες λογαριασμούς και όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα βρίσκεται σε μια κατάσταση σημαντικά καλύτερη από εκείνη άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι για την οικονομική σταθερότητα του ευρωχώρου στο σύνολό του ίσως έχουν επίδραση ορισμένε χώρε ακόμη και είναι μικρέ. Αλλά οπωσδήποτε οι κανόνε ισχύουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω αυτό να το ξέρουμε. όλε οι χώρε είναι ίσε. Σα uh, e Σας ευχαριστώ, η Άστριτ, για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Είχατε εδώ την ευκαιρία να μας υπενθυμίσετε τις επιφυλάξεις σας όσον αφορά την εισαγωγή ενός φόρου για τις ε, ε, συναλλαγές στην Ευρώπη παρόλο που το σώμα ε, ψήφισε την υποστήριξή του για τα μέτρα αυτά χωρίς να περιμένει τη, μια μελέτη επιπτώσεων. Θα ήθελα να ξεπεράσουμε λίγο τις αιτήσεις αρχής για να περάσουμε στην ουσία. Τι θα σήμαινε συγκεκριμένα η εισαγωγή ενός τέτοιου είδους φόρου μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα μόνο στο επίπεδο της ευρωομάδας. Οι χρηματοπιστικές ε, αγορές λειτουργούν έτσι που ε, ακόμα και ένας φόρος ενός δεκάτου ή εκατοστού ε, του 1% θα είχε επιπτώσεις στις συναλλαγές. Εσείς, αν συμφωνείτε, θα ε, προτείνατε μια άλλη μέθοδο ούτως ώστε το, ο τραπεζικός τομέας να συμβάλλει διαφορετικά στην οικονομική κατάσταση. Στην ε, εισαγωγή σας σημείωσα ότι χαιρετήσατε το γεγονός ότι η Κομισιόν μελετά την εισαγωγή κάποιων εισφορών τραπεζικών, bank levies. Υπάρχουν διαφόρων ειδών φόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Και πού προτείνεται να εφαρμοστεί αυτή η νέα τραπεζική εισφορά που προτείνει η Κομισιόν. Γιατί δεν απαντήσετε ξεκάθαρα στην ερώτηση της κυρίας Κράτσα όσον αφορά τον Σύμφωνο Ευρώ που υιοθετηθήκε στις 11 Μαρτίου κατόπιν πρόταση Γερμανίας και της Γαλλίας για την επιτάχυνση των ε, οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Και ακριβώς εδώ στις 15 ε, Μαρτίου ο Σόκλο Γιούγκερ, ο πρόεδρος της Ευρωμάδας, είπε ότι αυτό δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία και μάλιστα είπε ότι όλα αυτά ήδη υπάρχουν. Εσείς πραγματικά πώς κρίνετε αυτό το σύμφωνο, κύριε Πρόεδρε. Μπορείς να είναι πολύ κακό για το τίποτα ή είναι μια διαμάχη μεταξύ των πολιτικών υπευθύνων που δεν ε, αντέχουν να περνάνε στη δεύτερη γραμμή. εάν κατάλαβα καλά, δεν θέλετε να συγκεντρωθεί η προσοχή αυτή τη στιγμή στις οικονομικές πολιτικές ε, για να μην αποστραφούμε από το κύριο θέμα, δηλαδή το θέμα της διακυβέρνησης του ευρώ. Και εμείς ε, συμφωνούμε ότι αυτή, αυτή η δέσμη των έξι προτάσεων θα πρέπει να εξεταστεί τώρα και οπωσδήποτε μπορείτε να βασιστείτε σε εμά εδώ να σας υποστηρίξουμε στην κατεύθυνση αυτή. Εάν σας κατάλαβα καλά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρος Άστριτ. Ε, τρία λεπτά και 45 δευτερόλεπτα μίλησες. Merci ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Όσον αφορά το φόρο για τι ε, συναλλαγέ, πραγματικά επιβεβαιώνω ότι η θέση μα. ισχύει. Και αν υπάρχει ένα τέτοιο φόρο τελικά, θα πρέπει να εισαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλιώς θα οδηγούσε σε μια διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των ε, στον συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη και εκείνων που γίνονται στο υπόλοιπο του κόσμου. Όχι μόνο στη ΣΥΠΑ, γενικά στην Αυσία, στις αυσόμενες χώρες κλπ. Υπάρχει λοιπόν και ένα πρόβλημα. Νομίζω δικαίως ζητούμε να υπάρχουν ίσοι κανόνες όσον αφορά όλο το πεδίο αυτό που θα πρέπει να υπάρχουν σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια υπάρχει εδώ ε, κάποια δυνατότητα εφαρμογής αυτού του επίπεδου πεδίου παιδί σε, σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση η οποία δεν αναφέρεται σε αυτό καθ' το φόρο που θα πρέπει οπωσδήποτε προσεκτικά να εξεταστεί. Όσον αφορά το δεύτερο σας ερώτημα, θεωρούμε ότι θα ήταν καλό αυτές οι εισφορές, αυτά τα λέβη που εξετάζονται διάφορες χώρες, όχι όλες βέβαια. Υπάρχει διαφορά διαφοραστάσεις από τις διάφορες χώρες. Η ιδέα της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία αυτές οι εισφορές μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα, τα, μία, τα σημαντικά μου φαίνεται ότι είναι μία ευφύης ιδέα. Το σύμφωνο ευρώ νομίζω ότι κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Διάφορα αναφέρονται στο σύμφωνο αυτό που κινούνται πραγματικά προς την καλή κατεύθυνση και που συγκεκριμενοποιούν τις ε, διαφερόμενες κυβερνήσεις αυτό που εμείς συστήσαμε. Είπαμε λοιπόν ότι υπήρχε μια διακυβερνητική πτυχή στο σύμφωνο του ευρώ που θέλαμε να εγγραφεί στα κείμενα διακυβέρνησης που εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά στοιχεία του συμφένου αυτού του ευρώ που θεωρούμε ότι θα πρέπει να εισαχθούν κατά κάποιον τρόπο στην συνήθη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ίσως και του ίδιου του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβουλίου θα συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να εισαγάγει κάποια στοιχεία έχοντας τη συνέντευξη των κυβερνήσεων σε αυτό το τομέα. Είναι θετικό, κινείται προς την καλή κατεύθυνση και θα πρέπει όσο το δυνατόν να ενταχθεί στο στη συνήθη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Πρώτα σε ευχαριστώ. Ε, το επόμενο ρώτησε ΕΛΚ. Ο κύριος Νίτρας. E, bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Od kilku miesięcy stoi pan na... Είσαστε στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Συστηματικού Κινδύνου εδώ, του, της ομάδας δηλαδή για το κίνδυνο και θα ήθελα να σα υποβάλω κάποιε ερωτήσει όσον αφορά κάποιου από του κινδύνου που εξαιρεστήκαν από την ομάδα αυτή. Ίσως κάνουν δυνάμει κινδύνοι, πραγματικοί. Καταρχήν, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εδώ και πολλού μήνε εργαζόμαστε για να θέσουμε υπό έλεγχο τα ελλείμματα των προπολογισμών των κρατών μελών. Πολλοί ευρωβουλευτέ λένε όμω, ότι αυτή είναι η αρχή και τα πραγματικά προβλήματα ίσως είναι τελικά η χρέωση των οικογενειών. Και θα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι το σημερινό επίπεδο της χρέωσης που είναι συγκρίσιμη στα διάφορα κρατημέλη παρόλο που έχουν διαφορετικές πολιτικές και σε ορισμένε περιπτώσει κάποιε κυβερνήσει προσπαθούν να περιορίσουν τα χρέη αυτά των οικοκυριών, άλλες τα ενθαρρύνουν. Είναι αυτός ένα πραγματικό κίνδυνος, μια πραγματική απειλή. Δεύτερη ερώτηση. Όταν εξετάζουμε το διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, κάποια πειράματα σε εννέα κράτη-μελή... ολοκληρώθηκε εδώ. Δηλαδή ένα πείραμα θέλετε να υπολογιστούν ή να ανοίξουν ανεξάρτητα μία ε, Αυτό είναι ένα πείραμα που απέτυχε γιατί τα κράτη-μέλη θεωρήσαν ότι το να αν χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά θα οδηγούσε στην ε, μείωση του ελλείμματος. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση του προβλήματος αυτού, του πειράματος μάλλον αυτού. Κυρία Πρόεδρε, έχω μία δυσκολία. Την πρώτη ερώτηση ευθύνεται προς τον πρόεδρο μια, προς εμένα ως πρόεδρο μιας άλλη ομάδας και εδώ έχουμε ε, κάτι το τελείως διαφορετικό πρόεδρος ναι, το πρόβλημα είναι η Επιτροπή μου, όχι εσείς. Παρακαλώ. Θα ήταν καλό να σας παρουσιάσω ε, τις απόψεις αυτής της ομάδας σε, σε μια άλλη ειδική ακρόαση ίσως. Γιατί η συνθήκη είναι απόλυτα σαφή σε αυτό. Ότι δεν είναι η ίδια ομάδα, δεν μπορώ να μιλήσω ταυτόχρονα και για τις δύο αυτές ομάδε. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αφήσω κατά μέρο την πρώτη σα ερώτηση. Αλλά όποτε θέλετε μπορώ κάλλιτα να έρθω εδώ υπό την άλλη μου αυτή ιδιότητα και να σας απαντήσω. να έχουμε την σωστή επικοινωνία βάσει της νομοθεσίας που ισχύει. Uh, Α έρθω τώρα στην επόμενη ερώτηση που αναφερθήκατε στα συνταξιωτικά ταμεία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα της λογοδοσίας και της ε, ε τις λογιστικές πτυχές αυτής της υπόθεσης. Το ξέρω ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να τα μελετήσουν πάρα πολύ προσεκτικά και να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα και με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτό το τομέα. Αυτό που ζητούμε είναι ένα συνδυασμό των σωστών ε, αποφάσεων με κρίση δηλαδή και τους συνήθεις ε, κανόνες της ε, ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή, καμία, κανένα κράτος δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει το σύστημα με της βασικής κύριας σύνταξης για να το αντικαταστήσει από ένα σύστημα pay as you go. Ευχαριστώ. Ε, ο Μάρκους, ε, θα υποστείτε λίγο ακόμα την ομάδα του ΕΛΚ. Ε, ο Μάρκος Φέρμπερ, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και πάλι. Το φωτίστε από διάφορες πλευρές αυτό το θέμα. Θυμάμαι σε μία από τις τελευταίες συζητήσεις εδώ μιλήσαμε και για τις δραστηριότητες της Κεντρικής ε, Τράπεζας Ευρωπαϊκής που ε, αγόραζε κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Αυτό πώς αξιολογείται. Γιατί ε, τώρα σύμφωνα με αυτό το νέο μηχανισμό θα μπορείτε να αγοράζετε και στην πρωτογενή αγορά. Αυτό τώρα σημαίνει παραβίαση της ρήτρα μη διάσωσης ή γίνεται πάντα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συνθήκων. Ο πρωτογενή εννοώ τώρα, το, στην πρωτογενή αγώνα και όχι δευτερογενή. Βεβαίω είναι εφικτό, απαντά ο κύριο Τρίσε, ε, υπό την ευρωπαϊκή συνθήκη. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι αυτό είναι σύνομο. Εξ όσων γνωρίζω, ε, σε αυτό κατέλησαν οι νομικοί μας σύμβουλοι, οι δικηγόροι οι δικοί μας και του Συμβουλίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομική υπηρεσία. Θα έλεγα ότι ε, ήδη το πράττουμε αυτό για να βοηθήσουμε να αποκατασταθεί μια πιο φυσιολογική και σωστή λειτουργία του μηχανισμού μας μεταβίβασης στην νομισματική πολιτική. Μάλλον του, μεταβατικού μηχανισμού αυτό το καιρό, του προσωρινού. Και βεβαίως γίνεται αυτό και σύμφωνα με τη συνθήκη και επίσης φρονούμε ότι ο μηχανισμός σταθεροποίησης θα μπορούσε να το κάνει μόνος του αγοράζοντας κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Σας έχω πει ήδη και το είδαμε ότι η απόφαση που είναι καταρχήν των κυβερνήσεων αποφάσεις επέτρεψε να ε, ε, αγοράζουμε πλέον και κρατικά ομόλογα στην πρωτογενή αγορά, κάτι που δεν κάνουμε αυτόν τον καιρό καθόλου. Έχει αποφασιστεί επί της αρχής από τους κυβερνώντες, ακόμα δεν ισχύει στην πράξη. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τώρα τη Λίσα Φερέιρα να κάνει την ερώτησή της. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και πάλι για το νομισματικό διάλογο. Έχω δύο ερωτήσει εγώ. Η πρώτη έχει σχέση με τους μηχανισμούς ακριβώς σταθεροποίησης της ζώνης ευρώ που συνοδεύονται και από το δέσμι της ανταγωνιστικότητας και έρχονται να ενισχύσουν το θέμα αυτό της ε, διακρατικής διακυβέρνησης διακυβερνητικής αντί για την κοινοτική μέθοδο. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο έχει επεξεργαστεί μια δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση που να βασίζεται όμως στην κοινοτική μέθοδο, όχι στη διακυβερνητική. Αυτά τα δύο ε, συμφιλιώνονται και με ποιο τρόπο. Ερώτηση δεύτερη τώρα. Τα μέτρα που προτείνονται, βράχει πρόθεσμα, μπορεί να αποδειχθούν υπερβολικά. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μακροπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα θα γίνει η προσαρμογή όχι με ε, περικοπές μισθό στις χώρες που δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά βοηθώντας τις χώρες αυτές να γίνουν ανταγωνιστικές, γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι οικονομίες της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο σημείο Σε ό,τι αφορά τη ε, θεσμική μέθοδο, πώς θα στηθεί αυτός ο μηχανισμός σταθεροποίησης. Θα θέλαμε, όσο γίνεται, περισσότερο να μας υποστηρίξει το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν χωράει καμία αμφιβολία από αυτού. Είναι κάτι το οποίο είναι και πάει για δική μας θέση. Δεν θα σας εκπλήξει αυτό. Και δική σας φαντάζομαι. Εγώ έχω ακριβώς την ίδια παρατήρηση και για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Εκεί λέγουμε ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι πάρα πολύ καλά και θα πρέπει να ενσωματηθούν και στην οικονομική διακυβέρνηση που και εσείς συζητάτε αυτόν τον καιρό. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανταγωνιστικότητα, θα ήθελα να επαναλάβω το εξής. Τι έχει πολύ κρίσιμη σημασία κάθε οικονομία να λάβει πλήρως υπόψη της το γεγονός ότι εξασφαλίζουμε πλέον τη σταθερότητα των τιμών με έναν τρόπο εξαιρετικά σαφή, γιατί από την αρχή εξηγούμε ε, ότι το όριο αξιολόγησης το benchmark είναι χαμηλότερο από 2 και κοντά στο 2. Βέβαια υπάρχει και ονομαστική εξέλιξη κάποιων τιμών και ε, τη μονάδα του κόστους εργασίας. Είναι και αυτός ένας παράγον. Και όπως είπατε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την παραγωγικότητα και πώς αυτή προοδεύει. Και όπω είπαμε και ε, ήδη, όσο περισσότερο αυξάνεται η παραγωγικότητα, σε όλες τις οικονομίες, τόσο περισσότερο περιθώριο λιγμών δίνουμε για να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και ε, για οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όσο περισσότερο εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, τόσο περισσότερο τονώνουμε και τη σύγκληση μάλιστα θα σας έλεγα εντός της Ευρώπης και εντός της Ευρωζώνης. I'm ε, ε, ακούω γενικά για περικοπές μισθών για τις χώρες που έχουν απολέσει την ανταγωνιστικότητά τους. Έχει σημασία και αυτό, διότι αυτό σημαίνει ότι το μοναδιαίο ε, ε κόστος εργασίας θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Η Γερμανία είναι προφανές ότι αύξησε την ίδια της, την ε, ανταγωνιστικότητα με αύξηση της παραγωγικότητας και συγκράτηση του κόστους γενικά. Και αυτό επιτρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη μεγέθυνση της οικονομίας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πράγμα ε, που είναι ένα πολύ σημαντικός στόχος στις οικονομίες μας, όπου ακόμα είναι υψηλή, ε, υπερβολικά υψηλή η ανεργία. Ευχαριστώ. Ο Γκέι Μίτσελ τώρα. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε τη Κεντρική Τράπεζα, η Ιρλανδική κυβέρνηση αγνόησε μερικέ προειδοποιήσει και τη Κομισιόν και άλλων. Και οι ξένοι επενδυτέ και οι Ιρλανδοί επενδυτέ επένδυσαν σε τράπεζε, επειδή είχαν εύκολο κέρδο. Και η Κεντρική Τράπεζα εξακολούθησε να έχει χαμηλά επιτόκια, αλλά δεν έλαβε υπόψη τον πληθωρισμό λόγω των τιμών των ακινήτων. Ο Ιρλανδός φορολογούμενος τελικά ανέλαβε όλη την ευθύνη, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ευθύνης για χρέος που δεν ήταν δημόσιο χρέος αλλά ιδιωτικό χρέος. Εσείς και η Κεντρική Τράπεζα επενδύσατε σε Ιρλανδικές τράπεζες και ανακυκλώνεται και ανακυκλώνεται και ανακυκλώνεται κεφάλαιο. Δεν είναι καιρός να γίνει μόνιμη αυτή η επένδυση και η Κεντρική Τράπεζα να γίνει μέτοχος και όχι να είναι δανειστής σε αυτή τη σημαντική στιγμή για την Ιρλανδία και για την Ευρωζώνη την ίδια. Τι λέτε για αυτού του είδους την πρόταση. Απάντηση. Ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα πριν. Η νομισματική πολιτική είναι ένα δεδομένο. Είναι δεδομένο για όλες τις, ε, τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυξάνουμε τα επιτόκια, τα αυξήσαμε μάλλον το τέλος του 2005 παρά την συμβουλή 10 κυβερνήσεων 12 θεωρούσαμε ότι έπρεπε να αυξήσουμε τα επιτόκια για να εξασφαλίσουμε σταθερότητα των τιμών. Αρνηθήκαμε να μειώσουμε τα επιτόκια το 2004 στις αρχές με επιτόκια 2% τότε και άλλοι είχαν επιτόκια 1% αλλιενό σε, σε ανεπτυγμένε οικονομίε. Αρνηθήκαμε να μειώσουμε τα επιτόκια. Οι επικεφαλεί μεγάλων χωρών μας λέγανε να κάνουμε το αντίθετο. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν. Μπορείτε λοιπόν να πείτε, ναι είναι χαμηλά τα επιτόκια για την Ιρλανδία. είναι τα κατάλληλα επιτόκια για να εξασφαλιστεί σταθερότητα τιμών για την Ευρωζώνη. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε σε αυτό. Οι εθνικές πολιτικές πρέπει να το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Και να επηρεάζουν αντίστοιχα τα πράγματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες δυσκολίες στην συγκεκριμένη χώρα κάθε φορά. Η Κεντρική Τράπεζα είναι η κεντρική τράπεζα και ασκούμε την ευθύνη μας και το χρέος μας ως κεντρική τράπεζα. Όπως κάνουν και ζητάμε και από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω. Είμαστε κεντρική τράπεζα. Και βασική μας υποχρέωση είναι να δρούμε ως κεντρική τράπεζα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κατ' Έχουμε κάμποσο χρόνο αυτή τη φορά. Θα κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Και μετά θα περάσουμε στο Catch the Eye σύστημα. Για τα τεστ εντοχή των τραπεζών. Το έχουμε ξαναρωτήσει αυτό. Και ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνη και διαφάνειας. και μερικοί κεντρικοί τραπεζίτες φοβόνται όταν ξέραμε τα πάντα για τις τράπεζες θα είχαμε μια κρίση εμπιστοσύνη. Αλλά οι αγορές θέλουν να ξέρουν πώς έχει η κατάσταση με το εθνικό χρέος όσον αφορά τις τράπεζες στα βιβλία των τραπεζών και τι γίνεται με την έκθεση της κάθε τράπεζας. Γιατί έχουμε, ζούμε τόσο βαθιά την κρίση εθνικού χρέους και οι χώρες πρέπει αλληλέγγυα να στηρίζουν η μία την άλλη. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό θα, είχαμε μια γερμανική τραπεζική κρίση άρα και η Γερμανία έχει συμφέρον να βοηθήσει στη διαδικασία αυτή πράγμα το οποίο και κάνει. Δεν θα έπρεπε όμως τελικά να έχουμε περισσότερη διαφάνεια προς το μακροπρόθεσμο όφελος και των τραπεζών και των επενδυτών και όλων και το θέμα του εθνικού χρέους στα τραπεζικά κατάστοιχα ε, να λαμβάνεται σοβαρότερα υπόψη σε σχέση με τα τεστ αντοχής. Απάντηση. Ευχαριστώ. Από ό,τι θυμάμαι, στα προηγούμενα τεστ αντοχής ή κόπωσης, Τα χρεόγραφα που είχαν οι διάφορες τράπεζες στα βιβλία τους εγγεγραμμένα είχαν γίνει δημόσια. Είχαν δοθεί οι Άρα ένας παρατηρητής, ένας αναλυτής μπορούσε να κάνει τη δική του αξιολόγηση με βάση αυτά τα νούμερα. Αν και ο κανόνας λέει ότι το, τα βιβλία των τραπεζών δεν πρέπει να αξιολογείται ε, με βάση τους κανόνες μόνο της αγοράς. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την πλέον υπόψη την ονομαστική αξία. Επαναλαμβάνω, αυτό έχει αποφασιστεί και δεν θα παίξω εγώ το ρόλο του υπεύθυνου άλλων. Εμείς Ε, έχουμε κάνει ορισμένε μακροοικονομικές υποθέσεις για το ίδιο το, το, το στρες κόμποσης. Ο αρμόδιος φορέας όμως, το EBA, θα, θα, θα, αυτοί θα κρίνουν τι θα δημοσιεύσουν και τι όχι. Από ό,τι ξέρω, πρόθεσή τους, μάλλον, είναι να κάνουν όπως έκαναν και με τα πρώτα τεστ κόπωσης. Οι τράπεζες δηλαδή να δημοσιεύσουν τι έχουν στα βιβλία τους. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω αυτό. Υπάρχουν άλλοι που έχουν την ευθύνη γι' αυτό. Αυτό που έγινε στο παρελθόν, πιθανώς να ξαναποφασιστεί πάλι το ίδιο. Πρόεδρος, ερωτήσεις. Mm. Πολλοί συνάδελφοι, ο Γκέι πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την απάντησή του. Μία άλλη ερώτηση. Δέχεστε ότι είναι πρακτικά αδύνατο η Ιρλανδική κυβέρνηση να λύσει το δημοσιονομικό της πρόβλημα που κληρονόμησε και να επανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες ταυτοχρόνως. Αυτό δεν γίνεται. Είναι υπερβολικό να ζητηθεί από μία χώρα μέλος. Απάντηση. Όχι, όχι η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας τα τελευταία τρία χρόνια είναι δεδομένες οι αποφάσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την διεθνή κοινότητα, όχι μόνο από τις Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Η διεθνή κοινότητα το ενέκρινε. Είναι αναγκαίο το πρόγραμμα αυτό για την φερεγγιότητα της ίδιας της Ιρλανδίας. Δεν θέλω να κάνω άλλες υποθέσεις. με τις σοφές και κατάγγελες προσπάθειες της Ιρλανδίας, της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, σιγά σιγά θα ξανακερδίσουν την αξιοπιστία που απαιτείται. Εγώ από αυτό ξεκινάω. Ότι δηλαδή η Ιρλανδία μπορεί να το πετύχει και θα το πετύχει. Πρόεδρος Σιλβί. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Κάτι με προβληματίζει στον τρόπο με τον οποίο μερικοί πιστεύουν ότι και με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι κυβερνήσεις θα κρατήσουν το λόγο τους. Θα μου πείτε τι άλλο να ελπίζουμε. Εγώ τι να πω, βλέπω από τη μια μεριά έχω μια διάγνωση ότι δεν τήρησαν τα άρθρα, ορισμένε από αυτέ του Συμφόρου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και δεν έκανε ότι θα έπρεπε όσον αφορά τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Το comply or explain, μήπω συνεχιστεί, μήπω συνεχιστεί ο ένα να δίνει στον άλλον βραβεία καλή συμπεριφορά μεταξύ του. Πρόεδρο, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Το comply or explain δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Comply, συμμόρφωση, συμμόρφωση σε αυτό που σας ζητάει η Κομισιόν, η Επιτροπή να κάνετε. Αυτή είναι η έννοια με την πρόσφατη βελτίωσή της. Πρέπει να έχουμε την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, της ειδική πλειοψηφία. Να μην έχουμε το ίδιο σύστημα αποφάσεων με αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό που στην δική μας αργό λέμε περισσότερο αυτοματισμό στον έλεγχο και την εποπτεία. Ωστόσο, ωστόσο, θεωρώ ότι η σημερινή δυσκολία που είναι μεγάλη και την ξέρουν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπεύθυνοι Και γι' αυτό ζητάνε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ περισσότερο στο μέλλον από ό,τι στο παρελθόν. Το 2004 και 2005 μπορούσαμε ατιμόρυτα να λέμε ότι ο Σύμφωνος Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν μια ηλικιότητα, υπερορθόδοξη. Μερικοί έλεγαν την επέβαλαν ορισμένες χώρες που είναι υπερορθόδοξα, ενώ οι χώρες αυτές οι ίδιες προβληματιζόντουσαν σχετικά με το σύμφωνο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι δώσαμε μάχη η Κομισιόν και εμείς, η Κεντρική Τράπεζα, αντίθετα σε μια βούληση που ήθελε να το ακυρώσει το σύμφωνο αυτό και που οδήγησε σε μια νομική διαμάχη μεταξύ του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Δίκη, στο δικαστήριο φτάσανε τα δύο αυτά όργανα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο στεναροί στη διακυβέρνηση που ασκούμε και συμφωνώ με αυτό που είπατε. Εμπιστοσύνη μέχρι σε ένα ορισμένο βαθμό. Χρειαζόμαστε γερά θεσμικά όργανα στα οποία να έχουμε εμπιστοσύνη. Τόμας Μάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, πρόσφατα ε, ακούσατε στη Γερμανία να σας χαρακτηρίζουν ως Γερμανό-Γάλλο. Ε, βέβαια, ε, οι του συμφώνου σταθερότητα, ακόμα και αν οι χώρε μα δεν το τηρούσαν πάντα. Κάτι άλλο που δεχτήκατε επί κρίσης. Ε, εσείς πολύ μαζικά αγοράσατε ε, κρατικά ομόλογα, λέτε ότι είναι έκτακτο και πρέπει να κάνω μια κίνηση να στείλω ένα μήνυμα κατά των κερδοσκόπων. Εμείς όμως έχουμε κάποιες τράπεζες που θα πρέπει να εξασφαλίζουν κάποια συστήματα ε, που να τους προστατεύουν από κινδύνους. Αυτή η έκτακτη δαπάνη είναι κάτι το μεμονωμένο του παρελθόντος που τελείωσε ή θα πείτε ότι εάν ξανασυμβεί θα προσπαθήσω να αγοράσω αυτά τα περίεργα κρατικά ομόλογα για καλό σκοπό και το ξέρω και συμφωνώ για τη σταθερότητα των τιμών. Uh, Όπως σας είπα, αυτό που αποφασίσαμε ως τμήμα της νομισματικής μας πολιτικής είναι σε έκτακτες περιστάσεις να βοηθήσουμε να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός ε, στην παρακολούθηση της νομισματικής πολιτικής δεν είναι για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, είναι νομισματική πολιτική. Έχουμε κάποια στάνταρ μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για να παράγουν σταθερότητα και κάποια άλλα έκτακτα μέτρα ε, ε, ε, εφόσον η κρίση προκάλεσε κάποιες διαταραχές στις αγορές. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω και θα σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Η Ελίζα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να κάνω μια ερώτηση για αυτή τη διαδικασία ενίσχυσης ε, των τραπεζών και βοήθειας ε, και προστασίας από την πτώχευση σε περίοδους κρίσης. Μα ακριβώς είναι αυτή η μεγάλη πηγή κινδύνου να ε, έρχονται τα κράτη-μέλη να σώνουν τις τράπεζες. Δεν θα πρέπει να έχουμε κοινούς κανόνες και να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που να μας επιτρέπει να επιμεριζόμαστε ε, αυτό το άχθος σε περιπτώσεις πτώχευσης τραπεζών και να προστατεύουμε τους φορολογούμενους για να μην πληρώνουν φορολογούμενοι μία τράπεζα που πτωχεύει. Θεωρούσα ότι ε, ήταν δεδομένη αυτή η βούληση Τελικά τι έγινε, Εξαθμίστηκε, εξαφανίστηκε, γιατί στις αποφάσεις, τα συμπεράσματα της 11ης Μαρτίου λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης ότι η επέμβαση είναι υποχρεωτική και την αποφασίζει το εκάστοτε κράτος μέλος. Δηλαδή το κάθε κράτος θα πρέπει να δημιουργεί μηχανισμούς για να προστατεύει από τα προβλήματα πτώχευσης ενδεχομένως τραπεζών ή κρίσης τραπεζικής. Δηλαδή ο καθένας θα λύνει το πρόβλημά του σε εθνικό επίπεδο. Ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε λάβει μία απόφαση που έλεγε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το ζήτημα της κρίσης των τραπεζών. Ταυτόχρονα μιλούμε για κρατικά χρέη και για, για πτώχευση γενικότερα. Αλλά αποσιωπούμε το θέμα της πτώχευσης πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Απάντηση. Τα τεστ κόπωσης είναι ένας τρόπος ελέγχου της ε, ε των τραπεζών και ένας τρόπος ελέγχου αν κατά πόσον σε ειδικέ συνθήκες θα μπορούν να αντέξουν ή όχι. Δεν είναι για να εντοπίσουμε ποιοι είναι χρεοκοπημένοι και ποιοι όχι. Θέλουμε να δούμε τα επιπλέον στοιχεία, τις επιπλέον αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα, από τους μετόχους, από την ίδια την αγορά, αν χρειαστεί, ή εξαίρεση και από την δημόσιες αρχές για επανακεφαλοποίηση μιας τράπεζας στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν είναι επαρκώς κεφαλοποιημένη. Αυτό το προβλέπει φυσικά η κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει μηχανισμός επανακεφαλοποίησης τραπεζών αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της Ευρώπης. Έμεσα αυτό ζητήσατε. Είναι διαφορετικό αυτό από την έννοια του να έχουμε επίλυση ενός προβλήματος μιας ε, τράπεζα, α το πούμε, που καταραίει. Αλλά το εστρέ κόπο είναι το ίδιο. Και αυτό ισχύει και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ένα τρόπο ελέγχου να δούμε κατά πόσον είναι ε, οι τράπεζες ε, έχουν αυτή την ελαστικότητα προκειμένου ακριβώς να μην καταρρεύσουν. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για το εθνικό χρέος, η συμφωνημένη έννοια από όλε τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι μια έννοια που λέει ότι στην Ευρώπη θα έχουμε τον ίδιο ορισμό που έχουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το δόγμα εφαρμόζει το ΔΝΤ. Αυτό είναι. Και η υπόθεση είναι ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν θα χρεοκοπήσει. Έτσι ξεκινάει και το ΔΝΤ. Έτσι ξεκινάει και η Ευρώπη με αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η υπόθεση εργασία. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το νομισματικό διάλογο για σήμερα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τρισέ που είχε την αντοχή να χειριστεί και το σημερινό θέμα, ερωτήσεις, απαντήσεις και στο παρελθόν της συναντήσεις μας. Θα, θα δώσω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρο Μαργκάλιο γιατί θα πρέπει να πάμε τον πρόεδρο Τρισέ έξω για να μιλήσουμε στον τύπο μια σύντομη ανακοίνωση. Ακολουθεί το επόμενο σημείο της ημέρας διάταξη. Θα συζητήσουμε λοιπόν τις τροπο... την τροποποίηση των οδηγιών 2003 71 και την άλλη με ε, συγγητή τον κύριο Μπάλτ, στον οποίο δίνω μέσα στο λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στι 19 Ιανουαρίου τρέχοντο έτο, επιτέλου, επιτέλου τονίζω, μπόρεσα να αρχίσω την εργασία μου συγγητής ε, της ε, οδηγίας αυτής η Κομισιόν ε, είχε αναγγείλει και ξανά αναγγείλει ότι θα προετοίμαζε ένα πρόταση, αλλά δεν το έκανε. Είμαι άνθρωπο με υπομονή, αλλά δεν έχω πολύ κατανόηση ότι παρόλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που πέρασε, υπευλήθη ένα κείμενο ανώριμο, αν μπορώ να το πω έτσι. Ήδη το είπα αυτό προς την Κομισιόν. Έχουμε μια καλή σχέση εργασίας και γι' αυτό σήμερα δεν θα κάνω άλλες επικρίσεις. Η λεγόμενη οδηγία αυτή Omnibus 2 ε, είναι μια που αναφέρεται σε μια οδηγία πλαίσιο και στην οδηγία της συντάξης. Η τροποποιητική οδηγία χρειάστηκε ούτω ώστε να μπορέσουν οι διατάξει τη πτώχευση 2 στην συνθήκη της να προσαρμοστούν στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Στον τραπεζικό τομέα ήδη αυτό έχει εισαχθεί από την οδηγία Omnibus 1 του συναδέλφου Sanchez Προσέτ και ένα τμήμα μονάχα αναφέρεται στην Omnibus 2. Λοιπόν, όσον αφορά την οδηγία Omnibus 2, για να διευκρινώ κάπω τη συζήτηση, υπευλήθη ένα έγγραφο εργασία που το έχετε σήμερα μπροστά σα και το οποίο απεστείλει ήδη στα μέλη τη επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εγώ θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτό το κείμενο στην παρουσίασή μου. Ένα σημαντικό σημείο της Omnibus 2 είναι η προσαρμογή στη Λισαβόνα. Θα πρέπει να προσαρμοστούν οι διατάξεις στη συνθήκη αυτή. Η Επιτροπή το έχει κάνει αυτή τη λισαβονοποίηση, αν τη λέμε έτσι. Υπάρχουν βέβαια και πολλέ φορέ προσθήκε για τεχνικά εκτελεστικά πρότυπα. Φαίνεται όμω ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα τεχνικό τέτοιο πρότυπο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μέσω του κανονισμού για την Ευρώπη έχουμε δημιουργήσει μία νομική βάση ούτω ώστε η Ευρώπη να μπορεί να υποβάλει τεχνικά ε, πρότυπα διακανονισμού. Αλλά ενώ υπήρχε τα δυνατότητα δεν έγινε. Συμπεραίνω λοιπόν ότι όσον αφορά τις εκτελεστικές διατάξεις θα προσανατολισμούν στην Omnibus 1 και γι' αυτό η προθεσμία ε, επέμβαση του Κοινοβουλίου θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι τρεις μήνες και με μια παράτηση δύο μηνών. Είναι υποχρεωτική η διατησία μεταξύ των εθνικών ε, ε, υπηρεσιών. Υπάρχει εισαγωγή 12 άρθρων, ένα άρθρο το οποίο ε, αναφέρεται στο τέος, στη νέο επιτροπή ΣΕΟΠ, καθώς επίσης και σε άρθρα που δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τα άρθρα που μέχρι στιγμής είχε, είχαν συμμετοχή της ΣΕΟΠ της Ευρωπαϊκής Αυτής Αρχής η Κομισιόν κατά τη γνώμη μου, δεν έχει αντιμετωπίσει αυτό το σημείο. Η διαδικασία ε, σε όψη έχει αναγκαστεί από ε, μια διαδικασία ευρωπαϊκή και διαιτησίας. Αυτό σημαίνει απώλεια χρονική, ιδίως όταν ο παράγοντας χρόνος είναι πάρα πολύ στιγμή. Ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής κινητών αξιών και αγορών ε, είναι ένα θέμα στο οποίο θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε και άλλε παραδείγματο αυτή για τι ασφαλίσει που δεν συμπεριλαμβάνεται από την Κομισιόν ούτε στην 1 ούτε στην 2. Βέβαια θα υπάρχει και εδώ μια αναθεώρηση, αλλά δεν θα πρέπει εμεί να βασιστούμε στην επιβολή των χρονικών προθεσμιών τη Κομισιόν, αλλά θα μπορούσαμε έγκαιρα τώρα δηλαδή να αποστείλουμε κάποια μηνύματα. Αυτό είναι μια ανοιχτή σκέψη που θα ήθελα να συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή μας. από πολιτική απόψεω είναι πάρα πολύ σημαντική η Omnibus 2 όσον αφορά την ε, πτώχευση 2. Γιατί η Κομισιόν προτείνει ε, μία πρημοδότηση όταν ε, υπάρχει πίεση στην ρευστότητα της αγοράς. Εδώ εγώ θα το πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δεν θέλω να αξιολογήσω αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα ήδη τώρα να εκφράσω ότι χρειαζόμαστε μια εξασφαλισμένη βάση πληροφόρηση για να μπορέσουμε να εξτάσουμε το θέμα αυτό της πρημοδότηση ρευστότητα. Η Κομισιόν αναφέρεται επίσης στο διατακτικό, στο μελλοντικό διατακτικό, αλλά δεν επιτρέπεται αυτά τα τόσο σημαντικά τμήματα να ε, συγκεκριμενούν εκτός της οδηγία πλαίσιο και να μην υπόκεινε στην ε, λήψη απόφαση του Κοινοβουλίου. Το ίδιο ισχύει στην ε, στη στάνταρ μορφή που θα δώσει η Κομισιόν στο ΙΟΠΑ στο μέλλον. Στο ΙΟΠΑ λέγεται ότι θα πρέπει να μπορεί να αξιολογεί τις εξωτερικές ε, υπηρεσίες αξιολόγησης. Η Κομισιόν αναφέρεται στην οδηγία ιδίου κεφαλαίου. Αλλά εδώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρουσης με τον κανονισμό σε όπου αναφέρεται συγκεκριμένα για πρώτη φορά η δυνατότητα αξιολόγησης των ε, υπηρεσιών των εταιριών αξιολόγησης. Επίσης, υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, αξιολόγηση των τρίτων χωρών. Η Κομισιόν λέει ότι αν υπάρχει αρνητική αξιολόγηση για πέντε χρόνια, δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιπτώσει. Από αυτό ωφελούνται βέβαια οι ασφαλιστικέ εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι εξωτερικέ. Στι ευρωπαϊκέ εταιρείε η εξοικονόμηση κεφαλαίου είναι 50, λένε, δισεκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμόσουμε το άρθρο 227 και 260. Πώς μπορούμε να έχουμε εδώ ίσους ε, όρους ανταγωνισμού και τίθεται το θέμα του διεθνούς ε, πεδίου παιδής που θα πρέπει να είναι ισότιμο και δεν αναφέρεται επίσης τι θα μπορεί να γίνει μετά από τα πέντε χρόνια. Η δυνατότητα σύγκρουση, κύριε Πρόεδρε, ε, ενέχονται και οι μεταβατικές περίοδοι τρία ή δέκα χρόνια το πολύ. Η πρόταση Κομισιόν νομικά δεν είναι και πολύ εξασφαλισμένη. Κατά με αυτό που είναι σημαντικό είναι η πρωτης ε, κοινοβουλευτική αρμοδιότητα στην απόφαση και ελέγχου. Δεν επιτρέπεται η μέγιστη μεταβατική περίοδος να αναφέρεται στην ε, οδηγία αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει η συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη μεταβατική περίοδος, λέει η Κομισιόν, θα υπάρχει μόνο στο εκτελεστικό. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να πούμε παρά ναι ή όχι. Και αυτό ισχύει για όλο τη δέσμη εκτελεστικών διατάξεων. Εγώ συγχυτής θα εξετάσω πού χρειάζονται μεταβατικές διατάξεις και που θα μπορούμε να τις θέσουμε μέσα στην οδηγία πλαίσιο. Ελπίζω ότι έτσι η, ο, είναι χρήσιμη και η οδηγία της κρίς 5. Ορισμένα σημαντικά σημεία ε, τα έχω αφήσει κατά μέρο σήμερα, συμπεριλαμβάνονται όμως το έγγραφο εργασία. Θα ήθελα να πείσω στην προσοχή σας επίσης στο χρονοδιάγραμμα της Κομισιόν που υπάρχει στην πρώτη σελίδα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της ε, προθεσμίας εφαρμογής της Solvency 2. Εγώ δεν ξέρω γιατί να με καθυστερήσουμε, γιατί εάν η Κομισιόν ε, άρχισε τόσο πολύ να μας υποβάλει την πρόταση αυτή, γιατί εμείς θα πρέπει να βιαστούμε. Εγώ δεν θέλω να εθελοτυφλούμε ενώ του χρόνου για την Solvency 2, γιατί είμαι ρελιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να ακούσω τις αξιολογήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Βάλτ. Ο κύριος Σκίνερ. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη ταχεία απόκριση του, γιατί ξέρουμε ότι μας πιέζει ο χρόνος. Προφανώς ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να μελετήσουμε αυτή την οδηγία είναι δικός μας. Ε, θα πρέπει να μελετηθεί ε, σε βάθος, να ελεγχθεί Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, σε ό,τι αφορά τη φερεγγιότητα 2 και ως κληροδότημα της Omnibus 1 θέλουμε να διαδραματίσουν το σωστό ρόλο οι αρχές που μόλις τώρα ιδρύονται. Και πραγματικά θα πρέπει να ε, το ε, ε, μελετήσουμε με την ησυχία μας και συμφωνώ. Χρειάστηκαν 15 μήνες για να φτάσουμε ως εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι όταν συζητούμε αυτά τα θέματα έχει σημασία για τη φεραγγιότητα 2 όπως είπαμε αλλά και για την Omnibus 2. και η ίδια η οδηγία έχει τη δική της σημασία. Συμφωνώ όμως με τον εισηγητή είναι μάλλον τεχνικής φύσεως και λιγότερο πολιτικής. Τις λύσεις αναζητούμε και τις λεπτομέρειες τώρα, περισσότερο από ότι να εφεύρουμε νέα προβλήματα και να δημιουργήσουμε νέες ε, λύσεις για να παρακάψουμε την εφεργιότητα δύο που μπορεί ορισμένοι να ήθελαν. Ε, ορισμένα σημεία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και θα συζητήσουμε. Τα είπατε και εσείς κύριε Μπάλτς. Ε, δεν θα μπω Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των ε, πράξεων και των εφαρμοστικών διατάξεων και προδιαγραφών. Είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο να ε, εμβαθύνουμε και να αξιοποιήσουμε την εργασία που έχει ήδη κάνει ο κύριος Σάντσες Πρεσέντο. Και ξέρω ότι και εσείς ο ίδιος συμμετείχατε ε, δραστήρια. Ε, για το χρονοδιάγραμμα ε, δεν είναι μόνο κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα των μεταβατικών μέτρων γενικά και ε, ευρέως θα πρέπει να συζητηθούν. Παράδειγμα, υβριδικά μέσα. Στην ισχύουσα κείμενη ε, νομοθεσία, αρχικά προτανόταν 15 ετία, τώρα προτείνεται δεκαετία για τη εφαρμογή. Κάπου σε αυτό το χάος πρέπει να βάλουμε μία τάξη. Ε, για την ε, διατλαντική υπόθετο, μάλλον τις τρίτες χώρες και την παγκόσμια σύγκληση. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουν και οι τρίτες χώρες και ποια είναι τα αντίστοιχα εκεί. 54 ε, μέλη συν τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύσκολο να τις συντονίσεις. Και για τις εξουσίες μας, γενικά στο συμπέρασμα, Καταλαβαίνω προς τα που το πηγαίνει η καταλαβαίνω ότι θέλει να υπάρχουν πρότυπα, προδιαγραφές και να δοθεί σημασία σε θέματα πάρα πολύ κρίσιμα, ε, για τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε ε, μικρή πληροφόρηση. Ας πούμε το, το πριμ ε, ρευστότητας και άλλα θέματα που τα έχουμε συζητήσει στο, στο Solvency 2, αλλά ίσως όχι σε λεπτομέρειες, γιατί χρειάζεται να γίνει και διευκρίνηση και συζήτηση σε λεπτομέρειες. Θα έλεγα λοιπόν ότι το να ε, βασίζουμε την εργασία μας και σε ε, παραδοχές για υποθετικές τιμές ομολόγων τρομάζει τον κόσμο ε, για τα στοιχεία του ενεργητικού. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα γίνει συζήτηση. Εδώ χρειάζεται ένα μορατόριο να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα στο Solvency 2, ε, που τότε εκεί λύθηκαν. Δεν χρειάζεται να τα αφήσουμε αυτά τα προβλήματα τώρα να παρισπρίσουν στη σημερινή συζήτηση για τις equities πλέον. Τώρα, πώς θα γίνει η μεταφορά εξουσιών στην ΕΟΠΑ δεν έχω πρόβλημα να έχει τις εξουσίες που να μπορεί να χειριστεί. Γιατί το έχουμε συζητήσει και αυτό το θέμα της άμεσης εποπτείας και αν είναι πρακτικό που μπορούν να συμμετέχουν. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά, αλλά εφεραγγιότητα 2 είναι οδηγία και δεν είναι κανονισμός αφού βλέπουμε σιγά σιγά να αυξάνονται οι αρμοδιότητες που χωρούνται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σου ήθελε να το σχολιάσει και όπου θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να υπάρχουν αυτές τις εξουσίες στο μέλλον, όχι απαραίτητο τώρα, θα δούμε. Ε, να, ε, μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις γιατί δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ πόσο ε, σαφές είναι, πόσο απαραίτητο και χρήσιμο είναι να ε, κατακλειστεί και να συνθλιβεί η ΑΙΟΠΑ με υπερβολικές ε, αρμοδιότητες γιατί έχει έτσι κι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Κύριε Μπάλτς, πραγματικά κάνατε καταπληκτική δουλειά και σας ευχαριστώ. Η Σιλβί Γκουλά. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Να ευχαριστήσω τον Μπούρχαρτ. που μας έκανε το κείμενο, μας ετοίμασε το κείμενο αυτό πολύ σύντομα. Τον ευχαριστώ που ανέλαβε το θέμα αυτό και το έκανε με νυφαλιότητα. Επειδή Χρόνο πολύ δεν είχε και εμείς βέβαια σκεφτόμαστε παράλληλα στο χρόνο αυτό. Εμένα το κύριο πρόβλημά μου είναι να είμαστε ε, συνεπείς με αυτά που έχουμε στο πακέτο για την υποπτία. Να μην υπάρχουν ανακολουθίες. Αυτό βγαίνει από το έγγραφο εργασίας. όλες οι εκχωρημένες πράξεις λοιπά δεν είναι πράγματα που τα επινοούμε εξ αρχής, είναι δεδομένα αυτά. Από την άλλη μεριά πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμοστεί σωστά η Solvency 2, Solvency 2, 2. Μετά υπάρχει το νέο στοιχείο, ανάγκη για νέα απαιτήσει για τα νέα κεφάλαια για τις τράπεζες. Τι μπορούμε να ζητάμε δηλαδή από έναν ε, τομέα. Και μία ερώτηση. Αυτά που γίνονται στην Ιαπωνία θα έχουν επίπτωση σε ορισμένους ασφαλιστές επειδή οι καταστροφές είναι μεγάλες ακόμα καν δεν ξέρουμε το συνολικό τελικό νούμερο ορισμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πληγούν από αυτό ή όχι. Αυτό είναι ένα στοιχείο καινοτομία σε σχέση με το πακέτο εποπτεία. Ευχαριστούμε όμω και πάλι τον συνάδελφο ε, και για το αστόρα έργο και για τη συνεργασία. Φιλίπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Σιλβή είπε ότι επειδή έχουμε φως στην αίθουσα μας κάνει να είμαστε ε, να ακτινοβολούμε αγγελικά σχεδόν κάπως μια τέτοια έκφραση χρησιμοποιήθηση. Εγώ αντικαθιστώ τον Σβέν κάπως βιαστικά και επειδή δεν γνωρίζω πολύ καλά το θέμα γι' αυτό μπορώ να κάνω και μερικά λάθη. Πρώτον για το χρονοδιάγραμμα. Είναι θετικό το ότι έχουμε χρόνο γιατί το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να του δώσουμε το χρόνο που δικαιούται. Επειδή δεν είμαι ειδικό, ε, σας συγχαίρω για την σαφήνεια του κειμένου, συνάδελφε. Τώρα, μερικά στοιχεία που εμάς μας προβληματίζουν. Πρώτο, τις μεσολαβητικές εξουσίες της ΙΟΠΑ. Δεν θα θέλαμε αυτός ο κανονισμός Omnibus να χρησιμοποιηθεί για να ακυρώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις εξουσίες που δώσαμε στην ΑΙΟΠΑ με τον αντίστοιχο κανονισμό ίσα. Μη δημιουργήσουμε κερκόπορτες. Δεύτερο, κάτι που δεν το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν θέλουμε να δώσουμε ένα επιπλέον, χωρίς λόγο, άδικο, το πούμε, πλεονέκτημα στον ε, τραπεζικό κλάδο. Και αν εφαρμοστεί, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος, ας το πούμε, προφύλαξης, ώστε να μην έχουμε καταχρήσεις. Το επόμενο είναι, αφορά το άρθρο 260. Και αυτό δεν θέλουμε να αποτελέσει κερκόπορτα για να αποδυναμωθεί το μέτρο συνολικά. Και τέταρτο, μεταβατική περίοδος. Δεν έχουμε ακόμα το κείμενο της Κομισιόν, αλλά έχουμε το προηγούμενο κείμενο για τη Βασιλεία 3. Με ανησυχεί αρκετά το μεγάλο μήκος της μεταβατικής περίοδου. Το έχω ξαναπεί αυτό. Θέτε πόσο κυνηγάμε τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν χρεωθεί πάρα πολύ πόσο γρήγορα τους ζητάμε να βάλουν τάξη στα οικονομικά τους. Γιατί λοιπόν να έχουμε τόσο μεγάλη μεταβατική περίοδο για εταιρείε ή αξιολογητές κλπ. Ενώ ζητάμε από τις κυβερνήσεις να δράσουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν λέω να έχουμε το ίδιο μέτρο για όλους, αλλά να φροντίσουμε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό. Αυτό λοιπόν που μας προβληματίζει είναι μην τυχόν δώσουμε υπερβολικές εξουσίες να ορίσει την μεταβατική περίοδο, ενώ ξέρουμε ότι το λόμπι που ασκεί ο κλάδος αυτός είναι πανίσχυρο, στρέφεται προς την Κομισιόν πίσω από κλειστές πόρτες και είναι αποτελεσματική στη δράση τους. Αν θέλουμε να μειωθεί αυτό, και πρέπει να μειωθεί αυτού του είδους η δράση τους, θα πρέπει να παραμείνουν εξουσίες στο Ευρωκοινοβούλιο που να μας διασφαλίζουν ότι θα τους κρατήσουμε γραπωμένους στο αγκίστρε μας. Δεν είναι δουλειά της, των πολιτών και της κυβέρνησης. Μάλλον, αφού, επιτρέπουμε, αφού είμαστε δύσκολοι με τους πολίτες και με τις ε, κυβερνήσεις, γιατί να είμαστε ιδιαίτερα εύκολοι και επίοικείς με τον κλάδο αυτό. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Προηγουμένως όμως, επειδή έχω μερικούς επιζώντες από το Solvency 2, μερικοί από εμά που θεωρούμε ότι ξέρουμε τι κάνουμε και πριν και τώρα και μερικές από τις δεν μας βρίσκουν σύμφωνος δεν ξέρω αν ε, σωστά εντόπισε τους κακούς του παιχνιδιού, Φίλιπ, γιατί στη Solvency 2 υπήρχαν ορισμένοι άλλοι κακοί και μέσα στι χώρες μέλη και άσκησαν δράση λόμπι περισσότερο αυτοί παρά ο κλάδος στον οποίο αναφέρθηκες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ο καθένας να εκπροσωπεί τα συμφέροντά του, αλλά να ξέρουν ότι το ξέρουμε. Και τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή επίσης για το έγγραφο εργασίας του, το οποίο πράγματι με πολύ μεγάλη σαφήνεια περιγράφει τα θέματα της Omnibus 2, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής σας για τα σχόλια και τις ερωτήσεις να απαντήσω σύντομα. Πρώτο. για τον χρονικό ορίζοντα τη κατάθεση αυτή τη πρόθεση, καταλαβαίνω, γνωρίζω κύριε Μπάλτ, μιλήσατε για 15 μήνε. Ε, αυτό νομίζω είναι λίγο υπερβολικό. Κοιτάξτε, ήμασταν υποχρεωμένοι από νομική πλευρά να περιμένουμε να τελειώσει η Omnibus 1. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε την πρόθεση αρχικά να φέρει την πρόταση το Σεπτέμβριο. Βέβαια η συμφωνία για τη δέσμη ολόκληρη ήρθε αργότερα, γι' αυτό χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι να δημοσιευθεί ε, στην επίσημη εφημερίδα μέχρι να κάνουμε την πρόταση και από εκεί και πέρα να κάνουμε εμείς την πρόταση. Ε, είναι λίγο λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, από 15 μήνες και χαίρομαι που μπόρεσα να το διευκρινίσω. Στην ε, πρόταση αυτή θελήσαμε να ευθυγραμμιστούμε όσο γίνεται στην Omnibus 1 ε, και γι' αυτό το περιμέναμε γιατί ξέραμε ότι αν δεν το κάναμε, σωστά θα μας προσήπταν ότι βάλαμε ε, κάτι σε εφαρμογή για το τομέα των ασφαλιστικών εταιριών και για τις υπόλοιπες εταιρείε κάνουμε διαφορετική ε, προσέγγιση. Επίσης έγινε ένας λόγος για το πριμ ε, της έλλειψης ρευστότητας. Αυτό είναι λίγο σαν απομηχανής θεός ως έννοια στην πρόταση αυτή. Αλλά είναι τμήμα των συζητήσεων που έχουμε κάνει τους τελευταίους 15 μήνες ήδη με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους και αυτό το πριμ τι είναι. Είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε μετά τη χρηματοπιστωτική πίση. Ότι, σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν ένα παθητικό ε, συγκεκριμένο ε, δεσμευμένο, αλλά έχουν και ενεργητικό που μπορεί να είναι δεσμευμένο, γιατί είναι ε, ας πούμε προθεσμία ε, καταθέσεις και αυτό θα πρέπει επίσης να αξιολογείται, ότι μπορεί κάποιος να έχει ενεργητικό χωρίς ρευστότητα. Και στις εφαρμοστικές διατάξεις και μέτρα θα το δείτε εν ευθέτω χρόνο στην Επιτροπή σας αυτό κύριε Πρόεδρε. Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι εννοούμε. Σε αυτό το κείμενο δεν το έχουμε εντάξει διότι στις ασφάλειες έχουμε ενιαίους ομοιόμορφους κανόνες χάρη στο Κοινοβούλιο και στις προσπάθειές του και εσάς κύριε Πρόεδρε και πάλι θα ήθελα να ποτίσω ένα φόρο τιμής, ήταν δύσκολε οι διαπραγματεύσει, αλλά έχουμε λοιπόν ομοιόμορφους κανόνες για τις ασφαλιστικές εταιρείε, και αν κάτι πρέπει να αποφασιστεί αυτό θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακριβώς ε, αυτό ε, ο χώρος είναι η ΕΙΟΠΑ και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό ότι εκεί πρέπει να λαμβάνεται η απόφαση. Συμφωνώ κύριε Σκίνερ ότι δεν θα πρέπει να επαναδιαπραγματευόμαστε αυτό το θέμα της φερεγγιότητας 2. Φτάσαμε στο κρίς 5 που ήταν τεράστια επιτυχία, ε, πάρα πολύ μη. Δείχνει ότι είναι εφαρμόσιμο το σύστημα ε, Βεβαίω θα πρέπει ε, να οριστούν κάποια θέματα. Τώρα είναι πολύ νωρί ε, να αρχίσουμε την επαναδιαπραγμάτευση για τη φεραγιότητα 2 χωρί ακόμα να έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Στο ΚΡΙΣ 5, η τελευταία ποιοτική μελέτη σκοπιμότητας και αντικτύπου που μόλις ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε από την ΕΙΟΠΑ, θα συζητήσουμε τώρα με τους ενδιαφερμένους και με τα κρατημέλη τι συνέπειες πλέον και τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από τη μελέτη αυτή που ε, παρόδο είναι η μεγαλύτερη, ευρύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για, σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. 2.500 εταιρείε συμμετείχαν. Και ε, παρά αυτή την εξέταση θα φροντίσουμε και τα μεταβατικά στάδια. Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα φέρουμε κάποια στιγμή ένα κείμενο που θα ορίζει σαφώς ποια θα είναι αυτή η μεταβατική περίοδος. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει η σαφήνεια, η διαφάνεια για αυτά τα θέματα, αλλά όλα αυτά θα τα γνωρίζουμε μόλις μελετήσουμε τα στοιχεία της Κρίς 5. Έγινε λόγος επίσης για τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΙΟΠΑ και το τεράστιο άχθος με το οποίο την επιφορτίζουμε για να εκπονήσει δεσμευτικές προδιαγραφές. Τέλος του 2011 είναι ο χρονικός ορίζοντας. Νομίζω είναι τελείως ανεδαφικό αυτό και θα πρέπει να αναθεωρηθεί ήδη το συζητάει το Συμβούλιο. Θα χρειαστεί να ορίσουμε κάποιες προτεραιότητες. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι απολύτως απαραίτητο για την εφαρμογή της ε, Φεραγγιότητα 2 και τι μπορεί να αναπληθεί σε απότερο στάδιο. Για να οκληρώσω λοιπόν κυρία Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τα σχόλια του εισηγητού, ε, τα δικά σας σχόλια και τις ερωτήσεις στο μέλλον της Επιτροπής σας και προσβλέπουμε μαζί σας συνεργασία για να έχουμε μια πολύ καλή οδηγία Omnibus 2. Και επίσης θέλω να πω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως να μελετήσουμε το κείμενο και χαιρόμαστε γιατί το Φερεγιώτα 2 Solvency 2 είναι ένα τεράστιο εγχείρημα και ο κόσμος περιμένει την εφαρμογή του. Μιλάμε για πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και αν δεν μπορούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της 1 πρώτου 2013 ε, ε, θα είναι κρίσιμο. Αυτό το οφείλουμε στον κλάδο για όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βάλτς, θέλετε να ολοκληρώσετε. Ναι. Δεν θέλω να παρατείνω περιτά την συνεδρίαση γιατί έχει και ωραίο και ωραίο έξω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν και να τους ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Καραφακούλη για τις δικές του παρατηρήσεις. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια καλή και το κεντρικό μήνυμα που θα ήθελα να δώσω και να τονίσω σήμερα είναι ότι θα πρέπει πράγματι να ε, προσεγγίσουμε το θέμα αυτό τεχνικά και όχι πολιτικά. Εγώ συγητής ε, δεν ε, προτείνω να τροποποιηθούν οι διατάξεις του Solvency 2. Δεν ήθελα να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό τεχνικά και νομίζω ότι και οι σκιώδεις συζητητές, έτσι άκουσα τουλάχιστον, ε, θα είναι στο πλευρό μου. Χαίρομαι για τη συνεργασία των επόμενων εβδομάδων και αυτό ισχύει και τον Κάλ Φανκούλεν της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους συνεργάτες του. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πρώτη εταιρεία απόψε είναι πολύ καλή και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Thank uh, Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό ολοκληρώνει τις εργασίες μας για σήμερα. Μπορούμε να τελειώσουμε εδώ. Και θα σας δούμε αύριο το πρωί σε 9 για μια ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο Αλμούνια. Γεια σας.